So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήλθατε στη σημερινή μα συνεδρίαση τη Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, κυρία Τάισεν, την Επίτροπο που έχουμε καλέσει σήμερα στο σημείο 3 της ημερής σας ε, διάταξης, το πρώτο μέρος ε, του διαρθρωμένου διαλόγου μας όπου θα συζητηθεί το πρόγραμμα για το ε, τρέχον έτος. Θα επιθυμούσα να είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για τη συνομιλία με την ε, κυρία Επίτροπο. Ελπίζω να καταφέρουμε να κερδίσουμε ε, χρόνο σήμερα και μερικά λεπτά παραπάνω. Τώρα, καταρχάς, ε, ας περάσουμε στα διαδικαστικά. Νομίζω πως μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, πως δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Δεύτερον, Σήμερα δεν υπάρχει διερμηνία στα φιλανδικά, κροατικά και μαλτέζικα, δεν όχι, και ε, ιρλανδικά, μαλτέζικα έχουμε. Μετά έχουμε μία ομάδα επισκεπτών ε, προσκεκλημένων της ε, κυρίας Ούλφσκογκ, δέκα καλεσμένους από το Σουηδικό Συνδικάτο ΣΑΚΟ. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Έπειτα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την τελευταία συνάντηση ομάδας εργασίας σχετικά με την Ελλάδα. Στις 15 Μαρτίου ε, συνεδριάσαμε μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Συζητήσαμε πολλές λεπτομέρειες, ε, συζητήθηκε το θέμα της ανεργίας των νέων, της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως ε, καταλαβαίνετε και επίσης ένα θέμα που συζητήθηκε και είναι πάρα πολύ επίκαιρο και σοβαρό είναι η προσφυγική κρίση και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμβαθύναμε ε, στα, στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και αποφασίσαμε να συσταθεί μια νέα ομάδα παρακολούθησης την προηγούμενη εβδομάδα όμως μας ενημέρωσαν από την ε, ελληνική πλευρά ότι λόγω χρονοδιαγράμματος ε, θα ήταν καλό να αναβληθεί προγραμματισμένη επίσκεψη έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα για τις ε, συζητήσεις στα πλαίσια του Eurogroup. Γι' αυτό λοιπόν θα ορίσουμε νέα ημερομηνία για την επίσκεψη της ομάδας εργασία στην Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε αυτό την Πέμπτη κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Στο μεταξύ, Είχαμε και μία αντιπροσωπεία στην ε, Μπρατισλάβα ε, με ευκαιρία ε, της επερχόμενης προεδρίας. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εργασίας, Οικογένειας και Ευρωπαϊκών και Κοινωνικών Υποθέσεων και με τους ομολογούς τους εδώ. Συναντηθήκαμε με κοινωνικούς εταίρους, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αποκομίσαμε μια πρώτη εντύπωση για το τι προτίθεται να κάνει η Προεδρία της Σλοβακίας. Μετά, θα ασχοληθούμε με την εκστρατεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας κατά της δουλείας και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι σήμερα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης στις 6.30 το απόγευμα στον εξώστη θα διεξαχθεί μια εκδήλωση για, ε, την, ε, για μια νέα εκστρατεία του Παγκόσμου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας θα γίνει και συλλογή υπογραφών. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω σε αυτήν την εκδήλωση και να σας παρακαλέσω να παρευρεθείτε. Αυτά προς το παρόν. Στις 30 Μαΐου θα αλλάξει η ώρα συνεδρία τη Επιτροπή μα από τι 3.30 μέχρι τι 7 το απόγευμα. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί από τι 5 και μετά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τι υποχρεώσει μα και τα ταξίδια. Γι' αυτό λοιπόν, για να καταφέρουμε να τα προλάβουμε όλα, η Επιτροπή μα θα συνεδριάσει από τι 3.30 μέχρι τι 7. και στο διάστημα αυτό θα προλάβουμε να εξετάσουμε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία δεν θα αλλάξει. Αυτά λοιπόν όσα είχα να σας πω, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Αποτελεί τμήμα του διαρθρωμένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω, κυρία Επιτροπέ Τάισεν, θα πάρετε πρώτοι το λόγο, έπειτα οι σκιώδεις εισηγητές και μετά όσοι ήθιστε τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όταν παρουσίασα το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016 τον περασμένο Νοέμβριο, σας είπα ότι δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε συνήθως, ότι με την παρούσα συγκυρία πρέπει να βιαστούμε και να παράγουμε αποτελέσματα. Ε, δημοσιεύσαμε μία σύσταση για την καταπολέμηση της ε, μακρόχρονης ενεργείας, για το πώς θα φέρουμε τους ε, μακροχρόνια άνεργους ξανά στην αγορά εργασίας και πώς θα δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα για καταπολέμηση της αδύλωτης εργασίας. Σας ενημέρωσα επίσης για τις εξελίξεις στο δίκτυο έβρεσης εργασίας EURES. Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω ξανά, κύριε Μπερίνς και κύριε Μπέκερ, αρμόδιους ηγητές, για την εργασία σε αυτό το θέμα. Τώρα, από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενότητά μας έχει τεθεί ε, σε δοκιμασίες. Έχουμε περάσει πολλές δοκιμασίες από την προσφυγική κρίση μέχρι ε, την τρομοκρατία. Και αυτές οι συνεχιζόμενες προκλήσεις έχουν, ε, έχουν δοκιμάσει τον κοινωνικό ιστό και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν δείξει όμως ταυτόχρονα πόσο σημαντικό είναι να προωθήσουμε και να περασπιστούμε αυτές τις κοινέ αξίες. Ας εστιάσω τώρα στα κοινά θέματα τα οποία απαιτούν τη συνεργασία όλων μας. Καταρχάς, τα ευρωπαϊκά κοινωνικά δικαιώματα. Στις 8 Μαρτίου παρουσίασα στην Ολομέλεια μία πρόταση για έναν πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι η ουσία της ε, οικονομίας, της κοινωνικής η οικονομία της αγοράς είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα σε μια δυναμική οικονομία και ε, σε μια σύγχρονη κοινωνική προστασία. Οι οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πάντα σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτή η ισορροπία πρέπει πάντα να αποτελεί χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ένα μοντέλο το οποίο έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας, ένα μοντέλο το οποίο αποτελεί θεμελιώδες στατικό στοιχείο της ανάπτυξης και ε, δίνει ευκαιρίες σε όλους και λειτουργεί, ως, ε, και λειτουργεί ως οικονομικός σταθεροποιητής. Τώρα, αυτή η νέα κοινωνία που ε, χαρακτηρίζεται από καινοτόμα μοντέλα εργασίας και από αλλαγές έχει σημάνει την ώρα για να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και αν αυτό μπορεί να ταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Και οφείλουμε να αναρωτηθούμε εάν οι κοινωνικές πολιτικές μας στηρίζουν πραγματικά τους πολίτες, εάν ε, προστατεύονται από τους κινδύνους, εάν οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να ε, πραγματοποιήσουν όλες τους, ε, τις ε, δυνατότητες και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Όμως, όταν απαντούμε αυτές τις ερωτήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρέπει να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την αντοχή μας στις κρίσεις, ιδιαίτερα στην κρίση της Ευρωζώνης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία πηξίδα που να μας οδηγεί προς την ευρωπαϊκή σύγκληση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτή η πρόταση βρίσκεται σε στάδιο ευρείας διαβούλευσης συζητούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, διοργανώνουμε ένα διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων που, τις οποίες θα γυθεί ο κύριος Λάρσεν τον επόμενο μήνα. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό σας και με τη στήριξη που θα δώσει σε όλες τις εκδηλώσεις που ε, θα διοργανωθούν σε όλη ε, την Ευρώπη. Και ελπίζουμε το θέμα αυτό να συζητηθεί παντού σε κάθε χωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αυτή η συζήτηση έχει και διεθνές ε, βήμα. Συζητήθηκε στο Νταβός, στον ΟΣΑ και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας. Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την γενικότερη εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν ανυπομονώ να λάβω τα δικά σας σχόλια και τη δική σας, η δική σας συνεισφορά. Επίσης, στις 8 Μαΐου διατύπωσα την πρόταση για την αναθε... στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως για ορισμένους από εσάς αυτή η πρόταση ήταν ε, βιαστική και ε, υπερβολική, αλλά για άλλους ε, δεν έχει κάνει όσα έπρεπε. Δεν έχει φτάσει αρκετά ε, μακριά. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ και ε, κυρία Γιονχέριους, οι συνεισηγήτριες, είμαι σίγουρη πως θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, συζήτηση της πρότασης αυτής, εδώ όταν θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Αυτή η πρόταση έχει λάβει 14 αιτιολογημένες γνώμες από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα οποία ε, εκπροσωπούν ένα, την πλειοψηφία των, ε, των κρατών μελών. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να στηρίζουν την ενιαία αγορά και να συνεχίσουν να ε, στηρίζουν την ελεύθερη μετακίνηση με ίσους προς όλους κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται. Θεωρούμε την πρότασή μας αρκετά ισορροπημένη. Θεωρούμε πως είναι μια πρόταση που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, αλλά φυσικά θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις απόψεις όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, όσα μας έστειλαν. Έχουμε στη θέση μας όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα σχόλια που έγιναν. Τα σχόλια ήταν πολλά και διάφορα. Υπήρξαν ε, Πολλέ απόψει και αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούμε την ε, συνέχεια. Έπειτα υπάρχει και ε, το θέμα της προσβασιμότητας των ε, ατόμων με αναπηρία. Στην προηγούμενη Ολομέλεια σας ανακοίνωσα την πρόταση, το σχέδιο νόμου για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο και στο, στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου και από πλευρά Προεδρίας. Ακόμα τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει σε μια κοινή θέση, όμως μετά την πολιτική συμφωνία για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προσβασιμότητα στι ιστοσελίδε του Δημοσίου, είμαι πεπισμένη ότι στο Συμβούλιο οι Υπουργοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιτευχθεί συμφωνία στην, ε, για το θέμα της προσβασιμότητας. Επίσης, είναι πιστεύω σημαντικό η Επιτροπή Απασχόλησης να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για το θέμα αυτό και εδώ επαναλαμβάνω πως βρίσκομαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση ή όποια διευκρίνηση θέλετε. Σχετικά τώρα με τα άτομα με αναπηρία. Καλωσορίζω την έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία της Χέλγα Στίβεν για την εφαρμογή το, της σχετικά με τα άτομα με αναπηρία που συμπεριλαμβάνει και τις παρατηρήσεις ε, της ε, αντίστοιχης Επιτροπής των Ηνωμένων Επίσης, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η στρατηγική είχε καθυστερήσει κάπως γιατί αναμέναμε απαντήσεις ε, από τα κράτη-μέλη και από τους ενδιαφερόμενους φορείς στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Και μπορώ να σας πω ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα. Έχουμε την αναθεώρηση στη συνέχεια της ε, Οδηγίε για την επαγγελματική ε, υγεία και ασφάλεια και ξέρετε ότι εδώ ασχοληθήκαμε πολύ με τα λαξιογόνα. Είναι μία από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη. Τον ε, περασμένο χειμώνα σας ενημέρωσα ότι σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε και άλλους ουσίες ε, στον κατάλογο των καρκινογόνων και ε, μεταλλαξιογόνων ουσιών και στις 15 Μαΐου πριν από λίγες ημέρες ε, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και προτείνουμε αλλαγές σε αυτή την οδηγία για να περιορίσουμε ε, την έκθεση σε 13 καρκινογόνες ουσίες ε, στο χώρο εργασίας. Ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε λιγότερες περιπτώσεις ε, καρκίνου που εμφανίζεται στον τομέα της υγείας και ξέρετε ότι ο καρκίνος έχει μεγάλες συνέπειες ε, για το χώρο εργασίας, για τους πάσχοντες, για τις οικογένειές τους και την κοινωνία εν γέννη. Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί και μια επιπλέον ουσία, το κρυσταλλικό πυρίτιο, ε, κάποιες επιχειρήσεις έχουν καλό έλεγχο των αιωρούμενων συγκεντρώσεων αυτού του χημικού στοιχείου, ε, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι... Ε, αιτία και της ε, πνευμονοπάθειας λόγω του πυρητίου και ε, καρκίνου των πνευμόνων. Επομένως, ε, σκοπεύουμε να λάβουμε μέτρα για τον τομέα αυτό, διότι εκπροσωπούνται το 70% όλων των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυτό το κρυσταλλικό πυρίτιο. Ε, να σας ε, διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα σταματήσει εδώ το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε και νέους αναδυόμενους κυρδίνους και ε, θα προσαρμόζουμε και την νομοθεσία μας αναλόγως. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και είναι προτεραιότητα κάθε μέρα. Στη συνέχεια, ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής για εργαζόμενους γονείς ε, και άτομα τα οποία ασχολούνται με τη φροντίδα ε, άλλων ατόμων. Να ευχαριστήσω την κυρία Αρένα για την αφοσίωσή της στο θέμα αυτό. Σήμερα το πρωί είχατε μια ανταλλαγή απόψεων με την υπηρεσία μου και την Γενική Διεύθυνση Just ε, σε μια κοινή συνεδρίωση της Επιτροπής Γυναικών και Απασχόλησης. Ευπρόσδεκτη η πρότασή σας για την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να συγχαρώ και την εισηγήτρια, την κυρία Μπλινκεβιτσιούτε και την κυρία Τζανόκα και να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην ολοκλήρωση αυτής της ε, έκθεσης. Ξέρετε ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά από την απόρριψη της πρότασης για την ε, οδηγία ε, για την άδεια μητρότητας. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η οδηγία, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μια πρόταση η οποία έχει μπλοκαριστεί και δεν έχει καμία προοπτική να εγκριθεί, δεν μπορεί να συνεισφέρει σε τίποτα στη βελτίωση της ε, κατάστασης των εργαζομένων ε, γονέων. Ε, τώρα θέλουμε να προτείνουμε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που λαμβάνει υπόψη της και τις εξελίξεις και τις ανάγκες των σημερινών οικογενειών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να επιτύχουμε και το στόχο της προηγούμενης πρότασης, να άρουμε τα, ευρώ, τα εμπόδια για τη συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας, ανδρών και γυναικών και να υπάρχει κατάλληλη προστασία για εργαζόμενους γονείς. Ε, γονείς και άτομα που φροντίζουν ε, παιδιά και δαιμόνες ε, που δεν είναι γονείς. Αγαπητοί ευρωβουλευτές, όπως σας είπα στην εισαγωγή μου, η προσφυγική κρίση που συνεχίζεται έχει θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε δοκιμασία. Ε, υπάρχουν οι άμεσε ανάγκε των προσφύγων, αλλά πρέπει να προωθήσουμε επίσης και την ενεργό συμμετοχή τους στη χώρα υποδοχή, ιδίω στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία ενώ η αφομοίωση βεβαίως ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορούμε και εμείς να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να παρέχουμε και υποστήριξη και κίνητρα για τις δράσεις των κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να έχουμε καλύτερη ένταξη και να διευκολύνουμε και τη χρήση της απαραίτητης χρηματοδότησης ε, που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήδη επενδύει σε πολλά ε, προγράμματα ένταξη σε όλη την Ευρώπη. Και προκειμένου να διευκολύνουμε την ένταξη στην αγορά εργασία, πρέπει να προσφέρουμε μαθήματα γλώσσα, εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τα παιδιά και επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, πρέπει να επιταχύνουμε και την αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων τους και να διευκολύνουμε την πρόσβασή του στην αγορά εργασία. Οι πρόσφυγες ε, έχουν ποικιλία δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να συνεισφέρουν στις ε, οικονομίες μας ε, και στο μέλλον θα προτείνουμε και εργαλεία για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια στα προσόντα από τρίτες, ατόμων από τρίτες χώρες. Για να ολοκληρώσω για το θέμα αυτό, το κόστος της μη ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας θα υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της αντιμετώπισης οποιονδήποτε προκλήσεων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνολική απάντηση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα και να αποτελέσει και μια σημαντική ευκαιρία φυσικά αν τη διαχειριστούμε καταλήλους. Ε, κυρίες και κύριοι, Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω τώρα για το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες, το οποίο σας παρουσίασα με τον Επίτροπο Ναυράτσης πριν από ένα μήνα, ούτε θα σας πω περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο μόλις ε, περατώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την ε, ε, παρουσίαση των συστάσεων αναχώρα, μαζί με τον κύριο Ντομπρόσκη και τον Επίτροπο Μοσκοβισή θα σας παρουσιάσουμε το πακέτο στις 14 Ιουνίου, σε τρει εβδομάδες δηλαδή. Θα ολοκληρώσω λέγοντά σα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έκκληση για ανανέωση τη εταιρική σχέση μεταξύ κοινωνικών εταίρων και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ένα χρόνο αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι έδωσαν ε, τα καρπούς ε, αυτής της συνεργασίας μέσω πρόταση συγκεκριμένων δράσεων. Υπάρχει πρώτη διαβούλευση, όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 153 της Συνθήκης για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους τον Απρίλιο του 2015 και την ισορροπία οικογενειακής ε, και εργασιακής ζωής το 2015. Ε, όλα αυτά θα είναι η συνέχεια της δέσμευσής μας για τον κοινωνικό διάλογο, διότι όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ κάποια στιγμή, μπορούμε να έχουμε ε, μία αγορά εργασίας που να λειτουργεί όταν έχουμε έναν αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω με το εξή. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ υποσχέθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει κάποια πράγματα. Οι τομεί στους οποίους αναφέρθηκα, οι τομεί με τους οποίους ασχολείστε κι εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας ε, δίνοντα μεγάλα αποτελέσματα. Γι' αυτό ακριβώ και χρειαζόμαστε και την υποστήριξή σας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τι πρωτοβουλίες μας. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεχή στενή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θα αρχίσουμε τώρα με τον πρώτο γύρο συζητήσεων. Στην αρχή θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές, είτε οι, είτε αναπληρωματική του, Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον Τόμας Μαν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Πιστεύω πως κατέστη σαφές σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην ε, παρουσιαστούν ελλείψεις και προβλήματα. Έχουμε τις ε, δικές μας εμπειρίες από τις χώρες μας, οι οποίες όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων ε, έχουν τεράστιες διαφορές. Άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν, άλλοι δεν κάνουν τίποτα απολύτω. Και καταλαβαίνω όσους λένε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, ε, διότι υπάρχουν ελλείψεις. Από την άλλη όμως νομίζω πως πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία. Φυσικά και πρέπει να ε, φιλοξενήσουμε τους πρόσφυγες σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ε, φυσικά και δεν πρέπει να τους αφήσουμε μόνο στη μοίρα τους. Βέβαια, όταν ε, σίγουρα πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε η φιλοξενία των προσφύγων να είναι αξιοπρεπής. Από την άλλη όμως δεν πιστεύω πως ε, πρέπει να κάνουμε περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν υψηλό ε, επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ε, αλλάξει αυτό. και να προσέξουμε επίσης να μην ε, μεταφερθεί ένα πολιτικό ζήτημα στην ε, οικονομία. Η, στην Επιτροπή Απασχόλησης έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, αυτό το θέμα, όμως θα ήθελα να επαναλάβω ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, πρέπει να μείνουν μόνα τους. Ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες δεν πρέπει να τα αφήσουμε αβοήθητα. Ε, ας σκεφτούμε και τους ανθρώπους με αναπηρία που όπως είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αισθάνονται σε μειονεκτική θέση. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε δει τι γίνεται στη, Silicon Valley με την πρόοδο της τεχνολογίας και πόσο ε, ε, δύσκολος είναι ο ανταγωνισμός εκεί. Ε, κυρία Τάισεν, ξέρετε, πήγα πρόσφατα στι Ηνωμένε Πολιτείε, πήγα στο Πανεπιστήμιο του Μπέγκλε, συζήτησα με καθηγητέ εκεί και ξέρετε τι μου είπαν, ότι μακάρι να είχαμε και εδώ στι Ηνωμένε Πολιτείε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και αυτό είναι μια δουλειά η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό που χρειαζόμαστε, πιστεύω, εφόσον θέλουμε να λέμε πώ υπερασπιζόμαστε τα, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι να διατηρήσουμε με νύχια και με δόντια αυτό το μοντέλο που είναι τόσο αξιζήλευτο. Τέλος, όσον αφορά τους πρόσφυγες, πιστεύω πως είναι απαραίτητο να μάθουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία φιλοξενούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, μάθουν και να ενστερνιστούν έτσι και τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό που μας χαρακτηρίζει στην Ευρώπη, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσουμε να ενταχθούν οι πρόσφυγες πλήρως. Αυτό φυσικά δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αυτό χρειάζεται να γίνει βήμα-βήμα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Ευρώπη, αλλά από την άλλη πρέπει να φροντίσουμε αυτή η φιλοξενία να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρξει πλήρη ένταξη στην κοινωνία, έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσουμε και στους ε, πρόσφυγες τις ευρωπαϊκές ε, αξίες οι οποίοι μετά ενδεχομένω τις πάρουν στι ε, πατρίδε τους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εδώ να κάνω μια παράκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ζωάο Ροντρίγκε τώρα έχει το λόγο για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να αποτανθώ στην Επίτροπό μας, όχι μόνο ως πλήρες μέλος της Επιτροπής, αλλά και ως ε, η συντάκτρια για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμετωπίζει αυτή την μεγάλη κρίση που τα επικαλύπτει όλα. Ε, αν θέλετε όμως ε, μία, ε, μάλλον την ε, υποστήριξη των πολιτών, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα στον κοινωνικό τομέα, δηλαδή να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό ο ρόλος σας είναι ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. εκτιμούμε την εργασία σας από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας προσπαθήσατε να εξισορροπήσετε τους κοινωνικούς στόχους έτσι ώστε να υπάρχει σωστή αντιστάθμιση των οικονομικών μέτρων μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιταχύνατε την ε, ε, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας και αυτό μέσα στη, στα πλαίσια της απασχολησιμότητας και προτείνεται και ένα πακέτο κινητικότητας, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Χρειαζόμαστε όμως πιο ουσιώδη βήματα και γι' αυτό αυτή η συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι ύψης της σημασίας γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο και τα πρότυπά μας για να αντιμετωπίσουμε τις ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις σε σχέση δηλαδή με την ψηφιοποίηση, την ε, διαβίβαση πληροφοριών, τη, ιδιαίτερα την πρόθεση του τομέα της ενέργειας και όλα αυτά αποτελούν τη βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων από την άλλη πλευρά αντιμετωπίσουμε μία ε, κατάσταση, ανελισσόμενη κατάσταση η οποία υποσκάπτει τα κοινωνικά μας πρότυπα και αυτό αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωζώνης, κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τα κοινωνικά μας πρότυπα Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτός ο πυλώνας των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων να κινητοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να φτάσουμε σε μια κοινωνική σύγκληση στην Ευρωζώνη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία αλλά και για το μέλλον της Ευρωζώνης γιατί δεν είναι βιώσιμη η Ευρωζώνη μακροχρόνια εάν δεν έχουμε μία ανελισσόμενη κοινωνική σύγκληση. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πυλώνας θα πρέπει να οριστεί κατά τρόπον ώστε να ορίσουμε έναν κατάλογο κοινωνικών προδιαγραφών για ε, τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για όλους τους εργαζομένους. Ξέρουμε ότι ο, η τυπολογία της εργασίας αλλάζει λόγω της ε, ψηφιακής επανάστασης. Επίσης, θα πρέπει να μας απασχολήσει και η γύρανση του πληθυσμού, έτσι ώστε να έχουμε συστήματα προνοίας τα οποία να είναι βιώσιμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης ενός συστήματος είναι να αυξήσουμε το δίκτυο απασχολησιμότητας και αυτό είναι ύψης της σημασίας για τη βιωσιμότητα του κοινωνικού συστήματος. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τις δεξιότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαβίου κατάρτιση και αυτό με στα πλαίσια του εξισορροπημένου οικογενειακού ιστού για να μπορέσουν άντρες και γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, δηλαδή να ορίσουμε ένα ε, κοινωνικό πυλώνα ο οποίος θα εξισορροπήσει τα κοινωνικά δεδομένα. Δηλαδή ένας πυλώνας θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα ε, μέσα που να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Διαφορετικά δεν είναι πυλώνας. Και θα πρέπει να γίνει μια εξισορρόπηση σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της ΟΝΕ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας, αγαπητοί συντονιστές. Έχετε μόνο δύο λεπτά και ξέρετε πως είμαι γενναιόδωρος, αλλά όχι και τόσο γενναιόδωρος. Η Αντία Μάκιντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλά ευχαριστώ στη Μαρία Τάισεν για την σημερινή της παρουσία εδώ και για τις πληροφορίες που μόλις μας έδωσε. Και εγώ ανησυχώ εξίσου ότι εξακολουθούμε να διατηρούμε τα αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας και δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τα πράγματα και να, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν το 70% των θέσεων εργασίας θα μπορέσουν να το παρέχουν αυτό, να συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε ευημερία και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία. Δύο τομείς θα ήθελα να θίξω σήμερα. Ο πρώτος είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, την οποία έχετε σκοπό να κάνετε. Εσείς αναφερθήκατε στις αιτιολογημένες γνώμες και χαίρομαι που ε, σκοπεύετε να αξιολογήσετε τις αιτιολογημένες γνώμες που λάβατε. Με την εξαίρεση της Δανίας, οι χώρες ε, που ζήτησαν κίτρινη κάρτα, ε, μάλλον που δεν ζήτησαν κίτρινη κάρτα, είναι όλες οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει ενότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν θέλουμε να προτείνουμε μέτρα ή να προτείνουμε πράγματα που θα βάλουν τις ανατολικές χώρες ενώπιον των δυτικών. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της στα σχόλια και θα κατανοήσει τι ανησυχίες υπάρχουν πριν κάνει οτιδήποτε άλλο. Και κάτι άλλο από αυτού, το οποίο θα ήθελα να θίξω εν συντομία, είναι το εξής. Εγώ είμαι μεταξύ αρκετών που έλεγαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δούμε ε, πώς ε, εφαρμόζεται η εκτελεστική οδηγία πριν αρχίσουμε να αναθεωρούμε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Και η αντίθετη άποψη είναι ότι αυτά είναι άσχετα μεταξύ τους. Αλλά ακόμα και στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε αναφορά σε αυτήν την ε, αναθεώρηση ε, για την ενιαία ιστοσελίδα η οποία είναι τμήμα της οδηγίας του 2014. με ανησυχεί λίγο το γεγονό ότι βιαζόμαστε, ενώ εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να περιμένουμε. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω αφορά την αναθεώρηση του, του κεκτημένου και τι γίνεται, θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε στη διαδικασία και τι γίνεται με την ανοιχτή ε, ε, διαδικασία ε, η οποία είναι εξελίξη και με την ιδέα για καλύτερη νομοθεσία. Ε, τι κάνετε για να διασφαλίσετε ότι το ε, συμβούλιο το οποίο θα κάνει τον έλεγχο είναι πλήρες ε, αδέκαστο και αμερόληπτο. Τι μπορούμε να κάνουμε για την αναθεώρηση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Αναφερθήκατε σε αυτήν, αλλά φαίνεται να υπάρχει λίγη διαφάνεια και οι κοινωνικοί εταίροι δεν είδαν το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε τα σχόλια που έκανε το Ελεκτικό Συμβούλιο. Επομένως, ε, πώς ε, ε, συζητάτε με τους ενδιαφορομένους και την κοινωνία των πολιτών ώστε να μπορέσετε να αντλήσετε διδάγματα και να μπορέσουμε να έχουμε ένα νόμο με τον οποίο θα μπορεί κανείς εύκολα να συμμορφωθεί και να είναι και αποτελεσματικός. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ηλικιώτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να καλωσορίσουμε την κυρία Επίτροπο εδώ. Ε, αλλά πρέπει να δούμε πάντα τα δεδομένα και τα δεδομένα που έχουμε στη ζωή και να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα, μέχρι στιγμή βλέπουμε την Επιτροπή να μην πετυχαίνει κανέναν από του κύριου στόχου αναφορικά με τα ζητήματα απασχόληση και κοινωνική πολιτική για το 2016. Τα κράτη-μέλη δεν εμπιστεύονται την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, οδηγώντα τη σε κίτρινη κάρτα. Ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια για ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτά θα συζητηθούν στο πακέτο για την κινητικότητα, αυτό που βλέπουμε είναι συνεχώς να αναβάλλονται. Την ίδια ώρα η κοινωνική ένδυα και η κατρακύρα του κοινωνικού κράτους καλά κρατεί σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Στον Ευρωπαϊκό Νότο σχεδόν ένα στου τέσσερου Ευρωπαίου πολίτε, είναι το 24,6% με βάση τη στατιστική υπηρεσία, βρίσκονται στα όρια τη φτώχεια ενώ στατιστικά δεν δείχνουν και του τριγμούς στον πυρήνα της Ευρωζώνης και αναφέρομαι και στην ίδια τη Γερμανία με την ανεμική αύξηση των μισθών. Τέλος, η κοινωνικότητα των εργαζομένων μεταφράζεται πλέον σε υποχρεωτική μετανάστευση. Γιατί δεν μιλούμε για κινητικότητα, μιλούμε για κυρίω νέου ανθρώπου που αναγκάζονται λόγω τη ανεργία να μετακινούνται από τον Νότο ή την Ανατολή ε, προ τα κράτη που έχουν μια αναπτύξη. Εμεί ω αριστερά, ω Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, παραμένουμε προσιλωμένοι στι θέσει μα πω αφενό η οδηγία για του αποσπασμού εργαζομένου θα πρέπει να προωθεί την ίση αμοιβή για ίδια απασχόληση στο ίδιο μέρο, αλλά και να διασφαλίζει όλα τα κοινωνικά δικαιώματα των αποσπασμένων όπω αυτά καθορίζονται από το κράτο μέλο στο οποίο εργάζονται. Αφετέρου, η κινητικότητα εργαζομένων πρέπει να είναι άρρηκτα δεμένη με την κοινωνική του προστασία και την αξιοπρεπή εργασία. Συνεπώ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα απευθύνω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι πώ σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει όλα τα κοινωνικά δικαιώματα και την ίση αμοιβή των αποσπασμένων εργαζομένων την ίδια ώρα που θα λύσει το αδιέξοδο τη αναθεώρηση τη οδηγία. Και η δεύτερη είναι πώ σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει όλα τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα πλαίσια του πακέτου για την εργατική κινητικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Χίλια συγγνώμη θέλω να ζητήσω. Ε, δεν φταίτε εσείς, φταίω εγώ που, κύριε Χάρκιν που σας έφαγα τη σειρά, αλλά έχω τόσες σημειώσεις που με μπέρδεψαν. Μαρίαν Χάρκιν, λοιπόν, ε, κανονικά θα έπρεπε να έχετε το λόγο πριν τον κύριο Σιλικιώτη, αλλά παρακαλώ. Αρχίστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, νόμιζα πως ε, με αυτά που φοράω φαίνομαι πιο πολύ, αλλά μάλλον όχι. Καλώς ήλθατε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια από αυτά που είπατε. Μας μιλήσατε για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ε, εάν προστατεύονται αρκετά οι εργαζόμενοι, εάν είναι σε θέση να ταπεξέλθει στι ε, προκλήσεις. Έχουμε όλων των ε, ειδών της οικονομίες και γνωρίζουμε πως οι εργαζόμενοι είναι πολλές φορές άτυχοι και πολλέ φορέ ξεφεύγουν από την νομοθεσία και έρχονται σε άσχημη θέση. Υπάρχουν όμω πάρα πολλέ περιπτώσει εργαζόμενων οι οποίοι προσπαθούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, δεν έχουν καμία κοινωνική ασφάλιση, δεν έχουν ε, ε, σύνταξη και γι' αυτό λοιπόν αναγκάζονται να καταφύγουν σε τέτοιες μορφές εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτός ο κοινωνικός ε, πυλώνας θα προστατεύσει αυτούς τους εργαζόμενους, διότι οφείλει να προστατεύσει και αυτές τις ομάδες εργαζομένων. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας είναι οι ανισότητες. Οι ανισότητες δηλαδή ε, και πώς αυτές εμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει την ε, πράσινη βίβλο, να δει αν μπορεί να λάβει κάποιε αποφάσει και να εξάγει κάποια συμπεράσματα από αυτό. Μα μιλήσετε επίση για τη νέα ατζέντα για τι δεξιότητε. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν ένα σύντομο σχόλιο. Ε, εμείς θα επιθυμούσαμε ένα συντονισμένο διάλογο ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τους ε, φορείς της αγοράς εργασίας, δηλαδή τους φορείς ε, στον εκπαιδευτικό χώρο, τις επιχειρήσεις, για να δούμε τι γίνεται, ποια θα είναι η μελλοντική ζήτηση σε δεξιότητες και πώς θα συνδυαστεί η εκπαίδευση και οι δεξιότητες με τις θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και να υπάρξει συμφωνία, διότι πραγματικά χρειάζεται να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχει γίνει στην προσβασιμότητα, όπως αυτό που είπατε για την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες του Δημοσίου. Τέλος όπως είπατε, η νομοθεσία για κάποιους είναι υπερβολική και για κάποιους δεν είναι αρκετή. Έχω ρίξει μια ματιά στις διαφορές αντιρρήσεις των κρατών μελών και θεωρώ πως αυτές τις περισσότερες φορές βασίζονται σε αυτήν την υποχρεωτική ε, επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Για κάποια κράτη-μέλη αυτό είναι αρμοδιότητα εθνική και όχι ευρωπαϊκή. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, καλωσορίζει το γεγονός ότι θέλουμε ίση αμοιβή για ίση εργασία, όμως αυτό δεν είναι το ίδιο σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν φυσικά και άλλες αποχρώσεις σε όλα αυτά, αλλά με ενδιέφερε πολύ ε, να δω και την αντίθετη άποψη. Για παράδειγμα της Δανίας. Οι αμοιβέ, για παράδειγμα, θεωρούνται εθνική αρμοδιότητα, δεν συμπεριλαμβάνονται όμως στην αναθεωρημένη οδηγία. Εάν είχαν συμπεριληφθεί, αυτό θα έκανε διαφορά. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως το εξετάζει αυτό σαν, ένα, σαν μια πιθανή λύση Τέλος, συμφωνώ με την κυρία Μάκιντάιρ με το ότι παρά το γεγονός ότι συμφωνώ μαζί σας δεν μπορούμε να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάικελ για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ε, ήρθατε εδώ και προβήκαμε και σε μία σκόπιμη ανταλλαγή απόψεων στο παρελθόν, όπως γνωρίζετε. Θα ήθελα όμως να πω κάτι σε συνέχεια αυτών που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα σομβινισμό, ε, μία τάση προς ε, την εθνική ε, κυριαρχία και στην ουσία τι γίνεται, γίνεται ε, μία διάκριση κατά των μειονοτήτων, των κοινωνικών μειονοτήτων, των ε, Ρωμά, των προσφύγων, των μουσουλμάνων και ούτω καθεξής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει μια απάντηση σε αυτές τις ανισότητες. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος σας είναι ζωτικής ε, σημασίας. Χρειαζόμαστε δυναμικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμήσουμε αυτές τις ανισότητες. Θα ήθελα επίσης να μιλήσουμε και για τον κοινωνικό πυλώνα δεν μπορεί να είναι ένα συνονθήλευμα των όσων κάνουμε επί του παρόντος. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα όραμα για την τήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μία προστιθέμενη αξία στις ε, ευρωπαϊκές κοινωνίες και να αφήσουμε κανέναν πίσω. Νομίζω λοιπόν ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβαίνει σε αποκλεισμούς, όμως θα πρέπει να δώσετε μία όθηση και εσείς και άλλοι επίτροποι για να μην υπάρχει σοβινισμός και εθνικισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε σχέση με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ε, θα είναι μία από τις έντονες συζητήσεις μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Θα πρέπει να δώσετε φωνή όχι μόνο στα ε, εθνικά κοινοβούλια που υποστηρίζουν τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας, αλλά θα πρέπει να δώσουμε φωνή και στους εργαζόμενους που έτυχαν εκμετάλλευσης σε άλλες χώρες εξαιτίας των ελήψεων της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Επίσης, τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε, γιατί γίναν πολλές συζητήσεις για το πότε θα προωθεί το αυτή η συζήτηση. Από την ομάδα μου πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο ως προς την αγορά εργασίας. Τι θα κάνετε με την ατζέντα της πράσινης απασχόλησης. Έχετε ορισμένες γνώσεις ε, επί του θέματος. Το Κοινοβούλιο έκανε μια εξαιρετική εργασία. Θα δώσετε συνέχεια και αν ναι πώς. Ευχαριστώ πολύ. Λαόρα Τζά για το EFTD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε και πάλι. Μας ρωτήσατε αν το κοινωνικό μοντέλο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοντέλο κατάλληλο για τους πολίτες. Όχι, δεν είναι. Και η Ελλάδα αποτελεί μαρτυρία, εμβληματική ε, και προφανή ε, μαρτυρία ότι η, Ελλάδα, ε, ότι η Ευρώπη αποτυγχάνει παταγωγός τους κοινωνικούς της στόχους. 500.000 παιδιά σε απόλυτη φτώχεια στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει ούτε για αποτελεσματικό, ούτε για κατάλληλα μοντέλο. Ε, εδώ πρόκειται για μάχη επιβίωσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο σθένος και να πει λίγα λιγότερα λόγια. Διότι όταν εγώ ακούω να μιλάτε για ε, μία δέσμη συγκεκριμένων συστάσεων αναχώρα, η οποία προωθείται από τους συναδέλφους σας Ντομπρόφσκης, ε, Μοσκοβισή. Ε, φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί ξέρω τι περιμένει τις χώρες στη συνέχεια και τι τους αναλογεί. Διαρθρωτικές ε, ε μεταρρυθμίσεις, δάκρυα και, έμας, και αίμα που τους ε, ζητούν να προχωρήσουν και να αλλάξουν τα κοινωνικά πρότυπα και να φτάσουμε σε φτώχεια, σε επίπεδα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στην Ευρώπη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιμένω λοιπόν θαραλές επιλογές, επιλογές ιδιαίτερα σημαντικές, διότι αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος Γιούνκερ θέλει μεγάλα αποτελέσματα. Ο κύριος Γιούνκερ πρέπει να προσπαθήσει να κάνει μικρά αποτελεσματικά προγράμματα τα οποία να βγάλουν από την απόλυτη ένδια τα εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ήδη πρώτη ανάγκη. Αυτό είναι η δέσμευση που θα έπρεπε να αναλάβετε. Αυτό θα έπρεπε να είναι το δικό σα, αλλά και το δικό μα καθήκον. Ελπίζω λοιπόν μέχρι το τέλο τη θητεία μου, μέχρι το τέλο τη παρουσία μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να πούμε ότι επιτύχαμε αυτό το στόχο. Ας βγάλουμε από τη φτώχεια τους Ευρωπαίους πολίτες που σήμερα ζουν μέσα σε αυτήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο Τάισεν που προσήλθε εδώ σήμερα το απόγευμα για να μας μιλήσει για τις έξι προτεραιότητες μέσα στα πλαίσια του 16-17. Είναι δύσκολο να αντιταχθούμε σε κάτι τέτοιο. Όλοι θα συμφωνήσουμε στο ημικύκλιο. Θα πρέπει να δούμε ε, τα αμαία για να έχουν προσβασιμότητα παντού και η ασφάλεια για τους εργαζόμενους μας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές και σε ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στα πλαίσια αυτών των ε, οδηγιών. Και άκουσα ε, τέσσερα άλλα σημεία και χάρηκα που τα άκουσα. Μιλήσατε για την χάρτα των κοινωνικών δικαιωμάτων και τα κοινωνικά δικαιώματα και μιλήσατε για μία κοινωνική σύγκληση. Αυτό είναι απόλυτα ε, σαφές και στην ουσία είναι σαν να ε, προσπαθείτε να ανοίξετε μια ήδη ανοιγμένη πόρτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να υπάρξει σύγκληση τη στιγμή που όλοι χτυπάνε σε αυτή την ε, πόρτα. Νομίζω ότι θα κάνουμε μία εξουδετέρωση προς τα κάτω, δηλαδή μία θα έχουμε μία ε, εκτοτική τάση. Το είδαμε στην Ελλάδα και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτή την ε, συνεχόμενη ε, ένδια. Ήδη από το 1996 και μετά μιλάμε για την απόσπαση των εργαζομένων. Βλέπουμε όμως ότι η οδηγία αυτή οδήγησε σε συντρίμια. Μιλάτε για την εγγύηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών και είσαστε υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει και υπάρχει κοινωνικό dumping, στο οποίο είναι ανοιχτές όλες μας οι χώρες. Άρα καταδικάζεστε σε αποτυχία. Τώρα, ως προς την ε, ε, ισότητα ανδρών και γυναικών, και θα κάνω μια μικρή υπέρβαση, εδώ, Πρόεδρε, όπως και όλοι οι άλλοι. Εξαίρετα. Είπατε κατά της εκπαίδευσης των παιδιών, δηλαδή τα παιδιά τα κρατάει η μαμά, η γιαγιά, η θεία, η νονά, δηλαδή όποιος περνάει από το δρόμο, ε, θα πάρει και ένα παιδί, η αντάς, ε, η δική μας ε, πρόνοια ή οποιοδήποτε άλλος. Εξαίρετα, κυρία Επίτροπε, σε σχέση με την ένταξη των προσφύγων στην εργασία, μα έχουμε 25 εκατομμύρια ανέργους. Πού θα εντάξουμε και τους ε, πρόσφυγες. Εσείς στην ουσία ε, υποθάλπετε τον εθνικισμό και τον ε, υπέρμετορο πατριωτισμό και οδήγηστε πολύ μακριά. Μάλιστα. Με αυτήν την παρέμβαση ολοκληρώνεται ο κύκλος των συντονιστών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω στον επόμενο γύρο συντονιστών να παραμείνετε εντός των δύο λεπτών, όχι όπως τώρα. Τώρα, έχω 12 μέλη της Επιτροπής εδώ που έχουν ζητήσει το λόγο. Εάν μιλήσει ο καθένας σας δύο λεπτά, τότε θα, ε, θα φτάσουμε στα 24 και η κυρία Τάισεν θα έχει αρκετό χρόνο να απαντήσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λίζα Πεθμωρών Σαρτιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την υποστήριξή μας, κυρία Επίτροπε, για την εργασία σας. Είναι απόλυτα σαφές δεν οικοδομήσαμε την Ευρώπη από το κοινωνικό σκέλος, αλλά όλοι σήμερα θέλουμε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα για να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνική Ευρώπη. Αυτό ακριβώς επιθυμούν και οι συμπολίτες μας. Ε, μιλώντας για αυτή την στοχοθετημένη αναθεώρηση επί της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, συμμεριζόμαστε ένα στόχο και άκουσα πόσο οι πολιτικές ομάδες είναι υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, των εργαζομένων και της δημιουργίας ενός κοινωνικού βάθρου μέσα στα πλαίσια της οδηγίας αυτής ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Θα ήθελα αυτή η διαδικασία της κίτρινης κάρτας να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν και θα ήθελα να σας πω ότι σε επίπεδο κοινοβουλίου θα προωθήσουμε αυτή την εργασία θετικά και επικοδομητικά ανεξάρτητα από αυτή τη διαδικασία που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης έχουμε κινητοποιηθεί για την σύγκληση αυτή, για την κοινωνική σύγκληση, για την επίτευξη της και βεβαίως μετά από 20 χρόνια θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή την οδηγία, να την στοχοθετήσουμε και να την εξισορροπήσουμε. δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και ομάδων και θα ήθελα να λάβουμε υπόψη ότι ιστορικά και πολιτικά οι χώρες είχαν μία διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Θα πρέπει όμως να προωθήσουμε το δυναμικό χαρακτήρα των ΜΜΕ, διότι το 82% των θέσεων που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούνται από τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ. Μέσα στα δύο λεπτά έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είπατε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις της Επιτροπής, γιατί όλες αυτές οι, οι ανησυχίες τις οποίες προαναφερθήκατε προέρχονται από το γεγονός ότι το κοινωνικό, ο κοινωνικός πυλώνας θα αποτελέσει ευσεβή πόθο εάν δεν υπάρξει μία οριοθέτηση με καθορισμό οροφών. Αυτός ο κοινωνικός πυλώνας δεν μπορεί να σταθεί από μόνος του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο συνοχής. Διαφορετικά, οι οικονομικές πραγματικότητες που βλέπουμε στη, σε αυτή την ε, κίτρινη κάρτα θα αναπαραχθούν. Γι' αυτό, όπως είπε και η Μαρία Ζωάου Ροντρίγκε, θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δημιουργία απασχόλησης στις περιφέρειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Τώρα, σε σχέση με αυτή την πλατφόρμα στην οποία αναφερθήκατε, εγώ εργάστηκα και με τους ε, σκιώδεις και με την Επιτροπή. Από όσο γνωρίζω, στις 27 Μαΐου θα γίνει η πρώτη συνάντηση της πλατφόρμας. Όμως έχει δοθεί έμβαση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Μιλάμε για μία εξισορρόπηση έτσι ώστε να τραπεί η αδήλωτη σε δηλωμένη εργασία. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα έχει το πρόγραμμα εργασίας σε αυτή την ε, πλατφόρμα για να γίνει αυτή η δυτή παρέμβαση. Ε, έχω υπερβεί, ε, υπερεύει το χρόνο κατά ένα δευτερόλεπτο. Ναι, σχεδόν, σχεδόν το καταφέρετε με τα δύο λεπτά. Dank u wel, eh, voorzitter. Κύριε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου επί τη ευκαιρία, αφού υπάρχει δυνατότητα, να μιλήσω Ολλανδικά και να σας ε, ξεκινήσω την ε, παρέμβασή μου με μία είδηση στην εφημερίδα με τίτλο «Αν ο κόσμος θεωρεί τους κανόνες ε, άδικους, τότε η Ευρώπη θα βουλιάξει». Ο τίτλος αυτός είναι από μία συνέντευξη με την Επίτροπο που ήταν ε, στο Άμστερνταμ εχθέ, σήμερα είναι εδώ στις Βρυξέλλες και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Εάν ο κόσμος θεωρήσει ότι οι κανόνες είναι άδικοι, τότε ελοχεύει ο κίνδυνο ε, να μην υπάρχει υποστήριξη για την εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, μειωθεί και άλλο η εμπιστοσύνη των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώ και ε, εμείς, όταν λέω εμείς, ε, νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος αρκετών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι εργασίες για την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ε, είπατε ότι πρέπει να εξετάσετε τα σχόλια που έγιναν και να δείτε ε, τι απαντήσεις δόθηκαν από το κοινό σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να παραμείνει η πρόταση. Ελπίζω να γίνει αυτό, ελπίζω να συνεχιστεί η πρόταση, μπορεί να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά να την επεξεργαστούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό για τις αγορές εργασίας μας. Όταν υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται τους κανόνες και κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να ε, χρησιμοποιήσουν τα παραφυράκια που τους προσφέρει το σύστημα και να τους παρακάμψουν, ε, τότε σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχω χρόνο, το ξέρω, αλλά έχω μια ακόμα ερώτηση. Τι μπορώ να απαντήσω στους πολίτες που εργάζονται στις οδικές μεταφορές, που λένε ότι τι θα γίνει με τους ε, κανόνες περί μεταφορών τώρα. Μάλιστα, η κυρία ούτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, που δεχτήκατε να συμμετέχετε στην συνεδρίασή μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε συστάσεις για τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν επεσήμανε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις του 2013 για τις επενδύσεις ε, για τα παιδιά. Η παιδική φτώχεια αυξάνεται συνεχώς ε, στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και πλέον έχουμε 27 εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από τη φτώχεια. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να καταπολεμήσουν την παιδική φτώχεια. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να αναλύσετε το αίτημά μας, αίτημα το οποίο σας έχουμε υποβάλει επανειλημμένος για την εγγύηση για τα παιδιά, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέσο δηλαδή για την καταπολέμηση της παιδικής ένδυας. Τώρα που γίνεται αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο μέσο για τα παιδιά και επίσης θα υπάρχει και ε, συγκεκριμένος προϋπολογισμός σε αυτή την περίπτωση. Το Κοινοβούλιο σε αυτή τη θητεία, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη θητεία, πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα γιατί αλλιώς θα συνεχίσουν να υποφέρουν τα παιδιά. Δεύτερον, Αναφερθήκατε στο θέμα της ε, συμφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Σήμερα είχαμε μια κοινή συνεδρίαση Επιτροπής Απασχόλησης και Επιτροπής ε, Γυναικών. Ήταν πολύ καρποφόρες οι συζητήσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση αυτή. Έχω και την εξής ερώτηση. Πότε σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει το δεύτερο στάδιο των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους ε, για την συμφιλίωση οικογενειακής και ε, εργασιακής ζωής και τι σκοπεύεται να προτείνεται και τη δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις. Η κυρία Ρίκμαν. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές είπατε πως έχουμε διαφορετικά πρότυπα σχετικά με το μισθολογικό, με το εργασιακό δίκαιο και με την κοινωνική πρόνοια. Είμαι από την Αυστρία και όπως ξέρετε η χώρα μου έχει αρκετά υψηλά κοινωνικά πρότυπα. Τι γίνεται όμως με τους εργαζόμενους από μια γειτονική χώρα οι οποίοι ε, λαμβάνουν ένα μισθό ο οποίος βρίσκεται κάτω από το όριο των συλλογικών συμβάσεων όταν εκείνος δουλεύει στην Αυστρία. Τι συμβαίνει δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση ε, και τι συμβαίνει με την κοινωνική ασφάλιση όταν ε, εξαπατώνται οι εργαζόμενοι που εργάζονται διασυνοριακά. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα τέτοιας ε, απάτης και σίγουρα δεν είναι ούτε νόμιμα, ούτε σωστά. Όμως υπάρχει ελλειπής έλεγχος και ελλειπής εφαρμογή των σχετικών οδηγιών. Και μπορώ να σας αναφέρω και πολλά παραδείγματα τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απολύτως απαραίτητη μια μεταρρύθμιση της ε, νομοθεσίας διότι δεν γίνεται να ζούμε σε μια Ευρώπη όπου ένας ε, προσπαθεί να εξαπατήσει και να καταπιέσει τον άλλο και να ζούμε σε μια Ευρώπη που δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ελάχιστα κοινά πρότυπα. Και αντί να ε, διδασκόμαστε από τις βέλτιστες πρακτικές, προσπαθούμε να ε, εκμεταλλευτούμε ένα τον άλλο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ. στην πρώτη που τήρησε το χρονομιλίαση. Η κυρία Ρένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις διάφορες επεξηγήσεις. Επειδή πολλά ζητήματα εφήγησαν, θα ήθελα να μιλήσω για δύο ζητήματα. Μιλήσατε για μια σύγχρονη πολιτική προστασία. Συμμερίζομαι αυτά που είπε η κυρία Μπιλκετσούτε σε σχέση με την σύγχρονη προστασία, ε, κοινωνική προστασία. Μιλάμε όμως για την εγκατάλειψη 26 εκατομμυρίων παιδιών τι προτείνεται για αυτή την κοινωνική πρόνοια, κάτι το οποίο για έναν τομέα που είναι απαράδεκτο στην Ευρώπη ως προς τα ανήλικα παιδιά. Τώρα, ως προς την οδηγία για τους αποσπασμένους, δεν συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να περιμένουμε. Η οδηγία του 1996 δημιουργήθηκε για την προστασία των εργαζομένων και σήμερα χρησιμοποιείται για να γίνουν καταχρήσεις κατά των εργαζομένων. Δηλαδή έγινε μία στρέβλωση σε σχέση με την αρχική οδηγία. Θα πρέπει να την αλλάξουμε λοιπόν. Όχι κατά της κινητικότητας, αλλά υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να δεχθούν αυτήν την κινητικότητα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν χάσματα ε, αριστεράς-δεξιάς Ανατολής Δύσης. Θα πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Δεν θα πρέπει να υποπέσουμε σε καταστάσεις δουλεία στην εργασία, κάτι το οποίο ισχύει σήμερα στην Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο την εποχή μας. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Σάντερ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εργασία σας γιατί προσπαθείτε να εξορροπήσετε τον οικονομικό πυλώνα που είναι ισχυρός πυλώνας και της δημιουργίας αυτού του κοινωνικού βάθρου που αναμένουν όλοι οι συμπολίτες μας. Σας υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ένα ειδικό ζήτημα που σχετίζεται με μία γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε κατά δεύτερο μέρος της συνεδρίασης, δηλαδή ε, σε σχέση με την απασχόληση στις αγροτικές περιφέρειες. Ε, εκεί υπάρχει μία κρίση χωρίς ε, προηγούμενο με μία μεγάλη ένδια στα αγροτικά νοικοκυριά και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, κατά πόσο η Επιτροπή προβλέπει να εργαστεί για τις ε, κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην απασχόληση για να δούμε ποιες ε, εργασίες έχουν εξαρθρωθεί και τι επιπτώσεις υπάρχουν και στον αγροτικό τομέα αλλά και σε άλλους γιατί γνωρίζουμε ότι η εργασία στον, μία θέση εργασίας στον αγροτικό τομέα δημιουργεί πλήστες όσες σε άλλους. Αλλά νομίζω ότι τρεις, ε, είχαν άλλη σειρά πριν από σας, τρεις συνάδελφοι. Δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, Απευθύνομαι σε σας αλλά και σε όλους. Ακούσαμε τι είπε ε, ο κύριος Βάγνερ στην, για την Αυστρία, όπου χτες τις ε, προεδρικές εκλογές είδαμε ότι σχεδόν κέρδισε ένας εθνικιστής τις εκλογές. Μικρόφωνο. Ε, έκλεισε το μικρόφωνο σας. Ακούσαμε πόσο ο Ντομινίκ Μαρτέν ακούει τα, τις δικές μας αποστάσεις ε, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μπορεί να κερδίσει ο ένας ή ο άλλος. Ξέρουμε ότι υπάρχει η ελευθερία της μετακίνησης, υπάρχει η κοινωνική Ευρώπη που οδηγεί στην κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, θα πρέπει να επιτευχθεί με κοινούς κανόνες. Μιλάμε για κοινούς κοινωνικούς κανόνες, γιατί διαφορετικά δεν θα δεχτούν αυτή την κινητικότητα οι πολίτες. Σε σχέση ε, με τις προτάσεις σας που δεν πάνε πολύ μακριά, αλλά που θα πρέπει να μελετηθούν, θα ήθελα να εισακούσετε τους πάντες μέσα στα πλαίσια του γενικότερου συμφέροντος έτσι ώστε να μετακινηθεί η νομοθεσία και να προστατεύει τους κοινωνικά πιο ε, αδύναμους. Ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση και την εισαγωγή. Πρόκειται για μια συζήτηση που νομίζω ότι είχε πολλά ουσιαστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Θα πρέπει όμως να θυμηθούμε και τους κοινωνικούς εταίρους γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινήσαμε να ε, ασχολούμαστε εκ νέου με την αναθεώρηση τη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Στην αρχή σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετείχαν πλέρω οι κοινωνικοί εταίροι και για να υπάρχουν διαρκή αποτελέσματα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία στην οποία να μπορούμε να εμπλέξουμε και του κοινωνικού εταίρους. Εξακολουθεί να υπάρχει βέβαια δισταγμό από πλευρά κοινωνικών εταίρων, ιδίω όσον αφορά τα πιο περίπλοκα και ζητήματα, Επομένως, ε, προσπαθούμε να μην ε, δώσουμε αντίστοιχα παραδείγματα αυτής της μορφής, αλλά να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε τους πάντες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλές εξελίξεις στην αγορά εργασία. Όσον αφορά την οδηγία, την οποία αναφέρατε προηγουμένως ε, και η οποία σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας, είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει και πάλι ευθύ εξ αρχής να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι για να μπορούμε να έχουμε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Εμείς από πλευρά σοσιαλιστών και δημοκρατών θα υποστηρίξουμε όλες σας τις προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και εγώ μερικέ ερωτήσει. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ξανά που τοποθετηθήκατε κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ και όσον αφορά την ε, ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλάκις. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω όμως πώς ακριβώς ε, το βλέπετε, ποια ακριβώς είναι η άποψη που έχετε. Ένας Βέλγος δηλαδή που πηγαίνει να δουλέψει στην Ουγγαρία, τι συμβαίνει. Θα υπόκειται στην Ουγγρική εργασία και νομοθεσία ή όχι. Αν ας πούμε γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Ουγγαρία έχει ε, χαμηλότερους μισθούς από ότι το Βέλγιο. Ο Βέλγος λοιπόν εργαζόμενος ε, θα πρέπει να υπόκειται ε, στο, στις, στην Ουγγρική νομοθεσία ή όχι. Έπειτα, θεωρείτε πως το χρονοδιάγραμμα που μας αναφέρατε είναι εφικτό. Ε, ίσως, θα ήταν καλύτερο να μειωθεί ε, ο χρόνος σε έξι μήνες. έτσι ώστε να δούμε εάν τα κράτη-μέλη θα μπορούν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις και να εφαρμόσουν τους ε, κανόνες. Προβλέπεται επίσης κάποια ευελιξία σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και κοινωνική ασφάλεια έχετε κάποιες ιδέες για το πώς θα εξασφαλιστεί αυτό. Πώς θα είναι διαμορφωμένο, θα υπάρχουν κοινωνικές εισφορές. Τι θα γίνεται με την κοινωνική ασφάλιση, πού θα πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργαζόμενος, σε ποια χώρα αν είναι αποσπασμένος. υπό ποιε συνθήκες, υπό ποιε ρυθμίσει Έχετε κάποιες ιδέες γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γκουτιέρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φανταζόμαι ότι το γνωρίζετε, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που έχετε, διότι βλέποντας τα χθεσινά αποτελέσματα στις αυστριακές εκλογές, βλέποντας τι γίνεται με τα άκρα και τον λαϊκισμό σε όλη την Ευρώπη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας ελάχιστος κοινό παρανομαστής. Η μεγάλη αύξηση της ανεργίας, οι μεγάλες ανισότητες, η μεγάλη ε, σε ομάδες της κοινωνίας οι οποίες ε, αποκλείονται κοινωνικά και όλα αυτά έχουν έναν υπεύθυνο, το φόβο προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να αποστείλετε και ένα μήνυμα ελπίδες ακριβώς για να σταματήσει η αύξηση του λαϊκισμού και των ακραίων στοιχείων σε όλη την Ευρώπη. Και όταν αναφέρεστε στα προγράμματά σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις συστάσεις σας σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν κάποιες πολιτικές που τις θεωρούν ότι ε, τις προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ε, και εθνικές συστάσεις ε, για να σταματήσει ο κοινωνικός αποκλεισμό. Δεν υπάρχει κάτι για να σταματήσει η εργασιακή ένδυα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και ευρωπαϊκά προγράμματα για να σταματήσει ο λαϊκισμός και ο εξτρεμισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση ένα θέμα μεσοπρόθεσμο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και επιτροποί οι οποίοι προωθούν το εξή, ότι ένα πολίτη μπορεί να μεταφέρει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα, το ιδιωτικό του συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ε, με τη μία χώρα στην άλλη. Ε, μπορούμε να το κάνουμε όμω σε ευρωπαϊκή κλίμακα με τα δημόσια σχέδια ε, συνταξιοδότηση. Μπορεί να υπάρχει φορητότητα με τα κοινωνικά δικαιώματα. Μπορούμε να έχουμε μία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, στην οποία κάποιοι επίτροποι επιτρέπουν να μεταφέρονται ιδιωτικά ε, συνταξιοδοτικά συστήματα και δεν έχουμε ε, αντίστοιχα πράγματα για τα επιδόματα, για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τις συντάξεις ε, που δίνονται από το δημόσιο. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κυρία Επίτροπε, για μια ακόμη φορά μας περιγράψατε τι απόψει τη Επιτροπής σαν μέρος του διαρθωτικού διαλόγου. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δυστυχώς έχει αποτύχει πολύ απλά γιατί έχει επικρατήσει η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, του Βορρά και του Νότου. Η πρόοδο τη κοινωνία και ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων μόνο ως αστείο μπορεί να εκλειφθεί όσον αφορά την Ελλάδα. Πού είναι οι ίσες ευκαιρίε για όλου, πού είναι η αντίδραση των, των Ευρωπαίων στα επαχθή μέτρα που επιβάλλονται στην Ελλάδα, όλοι μιλάνε για αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη όμω επιλεκτικά. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο. Εντέχνω ο Υπουργό κ. Κατρούγκαλο απέφυγε να συναντήσει την, την αποστολή τη Επιτροπή μα με τη δικαιολογία ότι για τεχνικού λόγου αναβάλει τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι πω δεν έχει τι να μα πει. Η κυβέρνηση του ψήφισε απελευθέρωση απολύσεων, περικοπέ επιδομάτων, αύξηση του ΦΠΑ και τη φορολογία που όπω γνωρίζουμε όλοι μόνο ύφεση θα φέρουν και όχι την ανάπτυξη που περιμένουν. Το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν ούτε φάρμακο ούτε προσωπικό. Οι συνθήκε εργασία στα δημόσια νοσοκομεία είναι τριτοκοσμικέ. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση, η οποία τηρεί τι εντολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο ακέραιο, είναι οι δανειστέ να πάρουν τα χρήματά του. Όμω αυτά τα δανεικά δεν τα πήρε ούτε ο εργαζόμενο, ούτε ο μισθωτό, ούτε ο συνταξιούχο. Δυστυχώ, σε αυτέ τι κοινωνικέ ομάδε όμω έρχεται τώρα ο λογαριασμό. Θα μιλήσω για τους μετανάστες που έφυγαν από τη φωτιά του πολέμου και θέλετε να τους ενσωματώσετε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μα η ανεργία στις χώρες του Νότου καλπάζει. Παρακαλούν οι νέοι στην Ελλάδα για μια θέση έστω και χωρίς ασφάλιση, απλά για να μπορούν να επιβιώσουν. Εκεί δεν υπάρχει προστασία και τα πρόσφατα μέτρα θα φέρουν φτώχεια, περισσότερη ενεργεία και αδήλωτη εργασία. Όσο για τους συναδέρφους που ανησύχησαν για, τις, για την άναδο των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, να τους πληροφορήσω ότι τις βόμβες στις και στη Γαλλία δεν τις έβαλαν οι εθνικιστές, τις έβαλαν αυτοί που θέλετε να φέρετε τώρα στην Ευρώπη και να τους ενσωματώσετε. Ευχαριστώ. Τέλος η κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς την έκθεση για την εργασία. Ε, τι άποψη έχετε για την οδηγία σχετικά με την άδεια πατρότητας. Έπειτα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο κατάρτισης μιας προφορικής ερώτησης σχετικά με τη φτώχεια ε, και αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε σχέση με το μέσο εισόδημα. Η αρχική πρόταση στόχο είχε να φτάσει το κατώτατο κειμένο εισόδημα το 60% του μέσου εισοδήματος. Όμως δεδομένη της κατάστασης ε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο σκοπός στην ε, Λετωνία. Τη χώρα μου είναι κάτω το 50%. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο ξανά στην ε, κυρία Τάισεν, θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιε παρατηρήσει. Πρώτον, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνικά δικαιώματα. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχουμε συζητήσει και διαπραγματευτεί στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή, λοιπόν, συζητήσαμε το θέμα των ανισοτήτων στην Ευρώπη και έχουμε διαπιστώσει ότι, η μεγαλύτε... ότι έχουμε ε, τις μεγαλύτερες ανισότητες στην Ευρώπη από το 1961. Είναι, λοιπόν, έργο μας να ε, χτίσουμε ε, και να διορθώσουμε αυτές τις ε, ανισότητες όμως αμφιβάλλω αν θα καταφέρουμε να ε, έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε ε, Διότι οι πολίτες της Ευρώπης θα μας ρωτήσουν τι κάνουμε. Θα μας ρωτήσουν πώς μπορούμε να ε, εγγυηθούμε την ισότητα εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να, προστατεύει, που να τους προστατεύει. Δεν έχουμε απτά αποτελέσματα που να τα αισθάνονται οι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχίσουμε να βουλιάζουμε μέχρι ότου καταρρεύσουμε, μέχρι ότου η Ευρώπη από ε, μια Ευρώπη κοινωνικής επρόνοιας να καταστραφεί και να γίνει αγνώριστη. Έπειτα, ε, σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ήδη πως υπάρχει κατάφορη κατάχρηση της ε, νομοθεσίας και Ντανούτα με συγχωρείς αλλά ούτε και η οδηγία για την ε, επιβολή ε, αρκεί για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Δεν πρέπει να περιμένουμε διότι υπάρχει ο κίνδυνος τα κράτη-μέλη να υψώσουν ξανά τύχη. Έτσι ώστε de facto να αποτρέψουν την ελευθερία μετακίνησης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε ότι οι ορισμένε χώρε έχουν ήδη αρχίσει να ε, κάνουν κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε την οδηγία. Γιατί η αναμονή σημαίνει να πέσουμε στην ε, παγίδα αυτή που σας είπα και να υψώσουμε ξανά τύχη. Πιστεύω πως δεν αντέχουμε κάτι τέτοιο και ίσως θα ήταν μία λύση να προσπαθήσουμε να γκρεμίσουμε ε, αυτό, το, αυτό το τείχος που υπάρχει ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Ίσως θα έπρεπε στο Κοινοβούλιο προτού φτάσουμε σε ανοιχτή αντιπαράθεση, να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να γίνει μία άτυπη συνάντηση που, ε, στην οποία θα συζητηθούν όχι οι πολιτικές διαφορές, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια και να τα παραμερίσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια ε, σωστή λύση. Διότι θεωρώ απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να έρθουμε σε αυτήν την αντιπαράθεση από τη μία και από την άλλη να μην κάνουμε τίποτα το οποίο θα φέρει σε κίνδυνο αυτή ακριβώς την ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων. Αυτή η απραξία θα μας κοστίσει πολιτικά. Θα μας κοστίσει πολιτικά και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν ε, ως ε, παραπλευρά σχόλια. Θα δώσω τώρα αμέσως το λόγο στην κυρία Πίτροπο. Πρώτη ερώτηση κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις, τις οποίες σαφώς ε, θα λάβουμε υπόψη. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι πόσο χρόνο έχω. Αν μου δώσετε τρεις ώρες, εγώ να απαντάω τρεις ώρες. Σε 12 λεπτά θα τα καταφέρετε. Ε, εντάξει, 12 λεπτά. Συγγνώμη αν δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ε, διεξοδικά. Τα έχω σημειώσει όμως και θα τα λάβω υπόψη, πιστέψτε το. Αν μου επιτρέψετε θα απαντήσω στα Ολλανδικά γιατί είναι πιο εύκολο για μένα και να χρησιμοποιήσω και τις ε, πολύ καλές υπηρεσίες διερμηνίας που διαθέτεται. Όσον αφορά τους πρόσφυγες. Η ένταξη των προσφύγων πρέπει να γίνει καλύτερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα υπό την εξή έννοια. Ξέρουμε ότι όταν εξετάζουμε τις εκθέσεις αναχώρα, όταν εξετάζουμε την κατάσταση των μεταναστών στην αγορά εργασίας και την ένταξή τους στην κοινωνία, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι εξίσου επιτυχής η ένταξη. Πρέπει λοιπόν να γίνουν προσπάθειες. Υπάρχουν νέες αφήξεις στην κοινωνία μας, πρέπει να τους προσφέρουμε γλωσσικές δεξιότητες, να τους επιτρέψουμε να ενταχθούν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τους εκπαιδεύσουμε ε, ίσως και να τους βοηθήσουμε, ιδιαίτερα παιδιά που δεν έχουν ε, ε, ολοκληρώσει τη σχολική τους εκπαίδευση, να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας όπως έχουμε δεσμευθεί όλοι μας. Και φυσικά όλες αυτές οι προσπάθειες ε, μπορούν ε, να ε, καλυφθούν και από οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να προσφέρουμε επίσης και καθοδήγηση από τις υπηρεσίες μας. Υπάρχουν καλές εμπειρίες από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε όλοι και φυσικά ποτέ εις βάρος των πιο ευάλωτων πολιτών μας. Αυτό έπρεπε να το είχα πει ευθύ εξ αρχής. αν υπάρχουν αρνητικές προτεραιότητες για την δαπάνη ε, κονδυλίων, σίγουρα δεν θα πρέπει να γίνεται με ε, κονδύλια τα οποία προορίζονται για τους πιο ευάλωτους. Αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, ε, θα ήθελα να δηλώσω ευθαρσώς ότι έχουμε 507 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν όλοι συνεργαστούμε με καλό τρόπο και προσπαθήσουμε, θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε έναν αριθμό προσφύγων στις πολύ πιο πλούσιες κοινωνίες μας, αφού είμαστε μια πολύ πιο πλούσια περιοχή του κόσμου. Αν γίνει με έξυπνο τρόπο αυτό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Είναι ένα κόστος, βέβαια, θα χρειαστεί προσπάθεια και επένδυση σε νέο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά θα αποφέρει καρπούς. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν δημογραφικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτού του πράσφυγε ω τμήμα τη λύση και θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό το στοιχείο. Όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα. Σχόλια της κυρίας Ροντρίγκες. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που αναγνωρίζετε το έργο μας θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Αυτό ξεκίνησε από την επιθυμία μας να έχουμε ε, εκ των άνω σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προτιμούσαμε να είναι σύγκληση στην Ευρώπη των 28 και όχι μόνο στην Ευρωζώνη. Να έχουμε ε, εκ των άνω σύγκληση στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Νομισματική Ένωση, μια ένωση στην οποία υπάρχει το ίδιο νόμισμα, πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη ανταλλαγή κοινωνικών πολιτικών και αυτό είναι ε, απόλυτη ανάγκη, δεν είναι απλώς επιθυμία. Θα προτιμούσαμε βέβαια να εφαρμόζονται και στις 28 χώρες μέλη. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Θα ήθελα να σταθώ στη νομική μορφή του πυλώνα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τη συζήτηση. Ξέρετε ε, ότι θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό για να δούμε τι νομική μορφή θα προσλάβει ο πυλώνας αυτός, αλλά το σκεπτικό είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για δικαιώματα, αρχές και υποχρεώσεις δικαιώματα τα οποία ε, δεν θα πορέουν απαραίτητο από τον πυλώνα. Αυτή τη στιγμή θα καθορίσουμε αυτά, θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα προσαρμόσουμε την εργατική και κοινωνική πολιτική για τους πυλώνες αυτούς. Ε, τώρα, το κατά πόσο θα χρειαστούν και νομοθετικά μέτρα, ε, είναι κάτι ακόμα που πρέπει να εξετάσουμε. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν από νομικές πράξεις ε, στις οποίες υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είναι κάποια θέματα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα των κρατών μελών και μόνο και εκεί μπορούμε να έχουμε μόνο κάποια ορόσημα. Τα αποτελέσματα όμως της συζήτησης για το κοινωνικό πυλώνα δεν θα είναι απλώς μια σειρά από δικαιωμάτων που θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι ένα σημείο αναφοράς το οποίο θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, μπούσουλα για την πολιτική μας και από εκεί και πέρα θα δούμε ε, τις νομοθετικές προτάσεις που θα μπορέσαμε ίσως να προτείνουμε λόγω αυτού. Γενικότερα, και όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, ε, άφησα πάρα πολλέ ερωτήσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαράθεση Ανατολή-Δύση. Εάν υπάρχουν διαφορές, θέλουμε να τις περκεράσουμε. Είμαστε μια Ευρώπη 28 κρατών μελών, 507 ε, εκατομμυρίων κατοίκων και κατά την άποψή μας είναι όλοι ίσοι. Όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε με τις ε, τροποποίησεις είναι να είναι σαφέστεροι οι κανόνες. Θέλουμε να έχουμε δίκαιους κανόνες και να μπορούμε να τους εφαρμόσουμε στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν θέματα μισθών και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι υποχρεωτικοί κανόνες που ισχύουν για τους ε, ε, θα, ισχύουν και για τους αλλοδαπούς. Αυτή είναι η ουσία. Δεν θα παρέμβουμε στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι μισθοί στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία τέθησαν για αυτό το σκοπό. Ε, αυτό εξακολουθεί να παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πολύ συχνά οι κοινωνικοί εταίροι έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη διαπραγμάτευση των μισθών και φυσικά εμείς δεν θα ανακατευτούμε σε αυτό, δεν θα τα αγγίξουμε αυτό. Απλώς λέμε ότι οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν και που εφαρμόζονται για τους ε, εργαζόμενους σε μια χώρα θα πρέπει να γίνονται εξίσου σεβαστοί όσον αφορά τα επίπεδα των μισθών ε, ε, και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες βέβαια να το ξανασυζητήσουμε αυτό και στο μέλλον. Όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, Κυρία Μάκιντερ, εσείς ρωτήσατε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της προετοιμασίας. Οργανώνεται ένας πρώτος γύρος διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, επομένως ε, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Υπάρχουν αρκετές φήμες, ε, αλλά είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ακόμα οργανώνουμε την πρώτη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σίγουρα θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Και μετά είχαμε κάποιες ερωτήσεις περί ευελιξίας, ε, τι ζητάμε από τους εργαζομένους, νέες μορφές συμβάσεων, Ε, Πολλέ φορέ υπάρχουν συμβάσει αστικού δικαίου και όχι συμβάσει απασχόληση και θα, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ορισμένοι ε, άνθρωποι προστατεύονται πάρα πολύ καλά, κάποιοι άλλοι έχουν ελάχιστη προστασία. Δεν θα πρέπει οι άτυπε μορφές εργασία ε, να γίνουν κανόνα και κάποιοι άλλοι να απολαμβάνουν δικαιώματα και να προστατεύονται πλήρω και κάποιοι να είναι προστάτευτοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τομέα, Είναι τομέα στον οποίο ε, κάνουμε πολλά σχόλια στι εκθέσει εκθέσεις αναχώρα και στις συστάσεις αναχώρα. Επομένως μπορείτε να δείτε τις συστάσεις που κάναμε. Είναι κάτι που μας ανησυχεί και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση επί του θέματος. Όσον αφορά την ανισότητα, πρόκειται για κάτι το οποίο έχουμε προσέξει ιδιαίτερα και στις συστάσεις αναχώρα ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και από εκεί και πέρα επαφείται στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες, αλλά κάνουμε έκκληση να αντιμετωπίσουν τα θέματα της ανισότητας και μπορείτε να δείτε ότι είναι σαφέστατα εκπεφρασμένη αυτή η ανησυχία όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα. Για τις δεξιότητες, θα υπάρχει ένα νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες σύντομα και Μία από τι προτεραιότητές μα είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, με τους κοινωνικούς εταίρους και με τον ε, τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ε, για να διασφαλίσουμε ότι θα προετοιμάσουμε τους πολίτες καταλήλως για την αγορά εργασίας. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους ανθρώπους για την πραγματική ζωή, πρέπει να τους προσφέρουμε δεξιότητες, προσφέρ, ε, προσόντα, να τους μάθουμε αγωγή του πολίτη για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στην οικονομία. Πρέπει να έχουν και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τα πρώτα δηλάβηματά του στην αγορά εργασία και πρέπει φυσικά να αξιολογούμε και αυτές τις δεξιότητες, γι' αυτό ακριβώς και χρειαζόμαστε και την επιχειρηματική κοινότητα και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Προσβασιμότητα, η πράξη για την προσβασιμότητα. Για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των γυρεότητων πρέπει να σας συγχαρώ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευρά Κοινοβουλίου. Ε, με τα χαρά θα συμπεριλάβουμε και τις πτυχέ αυτές στην πράξη προσβασιμότητας και περιμένουμε και τη γνωμοδότηση που ε, θα καταρτήσει η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων για το θέμα αυτό. Να ξαναπεράσω στην απόσπαση των εργαζομένων. Οι αιτιολογημένε γνώμε που λάβαμε από τα διάφορα κοινοβούλια και οι επιστολέ σαφώς είναι στοιχεία τα οποία θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Θα αναλύσουμε προσεκτικά κάθε επιστολή, θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα σχόλια των Εθνικών Κοινοβουλίων και από εκεί και πέρα θα ε, συνταχθεί η απάντηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής και έχουμε διάφορα ε, ενδεχόμενα. Μπορούμε να την ε, προσαρμόσουμε, να την απορρίψουμε ε, ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Είναι μία λύση που θα αποφασιστεί επί τη βάση του περιεχομένου των επιστολών. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι ακόμα και πριν ξεκινήσει η πρόταση, εξετάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή τη επικουρικότητα. Πρόκειται για μια αρχή την οποία λαμβάνουμε πολύ, σοβαρή υπόψη, πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν είναι η υπόθεση ρουτίνα και θα πρέπει να γίνει σεβαστή επικουρικότητα. Αλλιώ δεν θα είχε γίνει πρόταση ούτω ή άλλω. Και πάλι όμω θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά τι επιστολέ, θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το ε, περιεχόμενο, θα απαντήσουμε και από εκεί και πέρα θα ε, ε, σας παρουσιάσουμε τη θέση μας. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε μια απόφαση. Δεν μπορώ να σας δώσω σαφή προθεσμία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναβάλλεται παόριστον. Πρέπει να διατυπώσουμε με μια απάντηση και ελπίζω να έχει γίνει αυτό πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιο είπε να λέμε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. στι συστάσει αναχώρα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα κοινωνικά θέματα. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή είναι η στάση αυτή της Επιτροπής. Μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες μόνο με αποτελέσματα και όχι με θεωρίες και ωραία λόγια και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κατάνουμε ό,τι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Επικεντρωνόμαστε στα θέματα στα οποία πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία ε, στα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα προκειμένου να δώσουμε καλύτερες δυνατότητε στους πολίτες ε, να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όλοι μα οι πολίτες. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να προσφέρουμε. Υπήρχαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων και των πολιτών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό προσών της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, γι' αυτό και ακριβώς θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την ελεύθερη μετακίνηση, την ελεύθερη κυκλοφορία και να μπορέσουμε να έχουμε μια ευθεντική εσωτερική αγορά που να είναι και έξι του ονόματός της. Ε, η εσωτερική αγορά δεν σημαίνει απλώς ανοίγουμε τα σύνορα και ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. Ε, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, συμφωνίες και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να εξετάζουμε τις προτάσεις μας για την απόσπαση των εργαζομένων. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα Ούτω ή άλλω αυτό κάνουμε και με το Συμβούλιο Υπουργών. Με κάθε ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε, εγώ ε, την εκμεταλλεύομαι. Προσπαθώ να μιλώ διμερό και με υπουργού από όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να επισημάνω το πρόβλημα τη απόσπαση των εργαζομένων. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με αποτελεσματικό τρόπο, βάσει στοιχείων, βάσει εξηγήσεων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται και να προσπαθήσουμε να βρούμε και κατάλληλε λύσει ε, μέσω διαλόγου. Αυτή είναι η μέθοδο μέθοδος που ακολουθούμε, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος και εγώ είμαι απόλυτα βέβαιη ότι ακόμα και σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα θα καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή απάντηση. Και τα δύσκολα γίνονται. Αν υπάρχει διάθεση, υπάρχει και τρόπος. Και αν υπάρχει και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπήρχε και μια ερώτηση για την πλατφόρμα ε, κατά της αδήλωτης εργασίας. και από όσο ελέγχθη αυτή η πλατφόρμα θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου, αυτά είπε και ο κύριος Πυρίνσκι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να φτάσουμε στη δική μας ατζέντα. Από όσο γνωρίζουμε θα υπάρξουν ε, πολύ ενδιαφερόμενοι επιθεωρητές από το χώρο της εργασίας και ζητήσαμε να ε, λάβουν υπόψη του τις διαφορετικές διαδικασίες επιθεώρησης έτσι ώστε να υπάρξουν ίδιες πρωτοβουλίες αλλά επίσης θα πρέπει όλες αυτές οι ιδέες και οι πρακτικές να συλλεχθούν έτσι ώστε να φτάσουμε σε συμπεράσματα που θα είναι πολύ καλά για την κατάρτιση πολιτικών και έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να καταρτήσει τη δική του ατζέντα. Και βασιζόμαστε σε εκείνους για να το κάνουν σε, κατά επικοδομητικό τρόπο. Σε σχέση με τη φτώχεια και τη φτώχεια των παιδιών, αυτό αποτελεί κάτι το επονίδιστο. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε και θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αλλά πρόκειται για ένα πολυσχηδές πρόβλημα. Δεν έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας στην Ευρώπη. Οι πολιτικές αρχές, τοπικές αρχές, οι περιφερειακές θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν μέσα στα πλαίσια του εξαμήνου Πολλοί είπαν ότι η απασχόληση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν θέλουμε δηλαδή να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες θα πρέπει να το κάνουμε μέσω της απασχόλησης. Θα θέλαμε να υπάρξουν ειδικέ συστάσεις στα κράτη-μέλη και αυτό ε, σημαίνει και ευελιξία και όταν ε, χρειάζεται υποστήριξη θα πρέπει οι πολίτες να έχουν ε, κοινωνική ασφάλεια. Και αυτό αφορά και την κοινωνική προστασία γενικότερα. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους ε, πολίτες να ανταποκριθούν και να μην μπουν στην παγίδα της ανεργίας. Εάν εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές στα κράτη-μέλη θα επιτελεστεί πρόοδος. Χαίρομαι ε, διότι το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχει προσδώσει μία ποσοστή αναλογία για την Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Και χαίρομαι γιατί τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις έτσι ώστε να κάνουν πολύ περισσότερα και αυτό το κατόφλι έχει ενταχθεί στο ΕΚΤ μετά από υπόδειξη του Κοινοβουλίου. Το δέχτηκε το Συμβούλιο και όπως ξέρετε ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα ζητήματα εις βάθος, κάτι το οποίο αποφασίστηκε πριν από δέκα ημέρες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή ε, εξισορρόπηση και στην ε, οικογενειακή ζωή. Θα θέλαμε μετά το θέμα της άδεια μητρότητας να κινηθούμε προς τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε τι θέλουν και εκείνοι. Θέλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία ή να την αφήσουν σε εμάς σε σχέση με την ε, παρεπόμενη αδιαπατρότητας. Εάν θέλουν αυτή την ευκαιρία θα τους τη δώσουμε. Θεωρούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ανταποκριθούν. Για τα, την πράσινη απασχόληση θέλουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση παντού, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην Ήπεθρο. Για άλλη μία φορά, λοιπόν, τα κοινωνικά δικαιώματα και η ελεύθερη κυκλοφορία συμβαδίζουν. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την, το κοινωνικό dumping και θα πρέπει να έχουμε έναν οργανωμένο επιχειρηματικό κόσμο στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Ε, η κυρία Στίβενς έθιξε το θέμα της οδηγίας για τους αποσπασμένους. Δεν έχω ε, χρόνο να απαντήσω, αλλά θα ήθελα να καταστήσω κάτι σαφές, γιατί υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Όταν λέμε ότι οι μισθοί και τα ημερομίσθια που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Μεδαπής θα πρέπει να ισχύουν και για τους αποσπασμένους, δεν σημαίνει ότι αυτός που έρχεται από μια χώρα που έχει ψηλότερους μισθούς θα κερδίσει λιγότερα. Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Και αυτό που είναι δύσκολο είναι το εξής. Οι αποσπασμένοι έχουν μία σύμβαση με τον εργοδότη από τη χώρα από την οποία προέρχονται. Αλλά εάν υπάρξει μεταφορά απόσπαση σε μία άλλη χώρα, όπου η μισθή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη, θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση με αυτή που ισχύει στην χώρα εργασίας, έτσι ώστε τα χρήματα που καταβάλλονται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εργαζόμενος έχει μία σύμβαση ε, από τη χώρα προέλευσης, με τη χώρα προέλευσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί και στη χώρα υποδοχής. Σε σχέση με το 60% το επίπεδο φτώχειας, θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε με ένα ε, μέσο εισόδημα που να ανταποκρίνεται στο 60%. Όπως ξέρετε, εμεί κάνουμε συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε ένα μέσο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω, Πρόεδρε, να μπόρεσα να θίξω έστω και επιφανειακά τα επιμέρους ζητήματα. Θα τα δούμε αυτά τα ζητήματα εις βάθος και σε επίπεδο Επιτροπής, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είχα ε, χρόνο να ανταποκριθώ πλήρως ε, στις ερωτήσεις σας και να τις απαντήσω πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε σχεδόν 12 λεπτά. Μας έμειναν κανένα πρόβλημα. Το ξέρω, το ξέρω, ποτέ δεν έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Και την επόμενη φορά θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 15 λεπτά και να προσπαθήσουμε, εάν οι συντονιστές μείνουν εντός ε, χρόνου ομιλίας, να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τώρα δεν τελειώσαμε εμείς δεν έχουμε τελειώσει ούτε με τον ε, διαρθρωμένο διάλογο. Αυτή τη στιγμή ε, εργαζόμαστε πάνω στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία θα συζητηθεί στις 26 Μαΐου ξανά στη συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουμε συμβαστικές προτάσεις να συζητήσουμε. Στις 30 του μήνα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και αν δεν υπάρξει συνένεση με τους συντονιστές, τότε θα ε, αν υπάρξει μάλλον συνένεση, θα, θα πάει στην διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών, μετά στη διάσκεψη των Προέδρων και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις δικές μας προτάσεις, τα δικά μας σχόλια και την κριτική στο πρόγραμμα εργασίας της για το επόμενο έτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα περάσουμε στις ψηφοφορίες.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 4, περνάμε στις ψηφοφορίες για τη νέα μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο Γιώχημ Σούστερ είναι εισηγητής. Έχετε μπροστά σας τον κατάλογο της ψηφοφορίας και αρχίζουμε αμέσως. Συμβαστική Β παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ? με ανάταση του χειρός. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Μ μη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Θα ψηφιστεί μαζί με την συμβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 32. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Συμβιβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Να στο το δούμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 64, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε, πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. Ε, J, υπέρ, κατά. Αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Τροπολογία 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Πώς είπατε παρακαλώ. Ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά το είδα. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 104. Άρα λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 42 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μάλιστα. Παίρναμε τώρα στο σημείο 5. Με ποιου τρόπου μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβαστική σε. Βιάστηκα, λέει ο πρόεδρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 και 37. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίθηκε. Θα θέλετε να το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 56. Πέρας. 34 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογής 59 και 60 υπέρ, κατά, αποχές Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε την 59 μόνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Όχι, όχι, δεν είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία. Έχει αποσυρθεί αυτή η πρόταση. Όλη την 70 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εβδομήντα ένα. Υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Εδώ έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται το πρώτο τμήμα, άρα καταπίπτει το δεύτερο. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 74, πρώτο τμήμα. Μάλιστα, 25 προς 25. Απορρίπτεται. Όχι, θα ψηφίσουμε και για το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Πολύ ωραία. 75. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 75. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. για την 90. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε και αυτό ηλεκτρονικά. 99. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 και 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική εν, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 124 και 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική όμικρον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. 6. Αξιολόγηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία 2013-2015. Συμβιβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 14. Άρχεται. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να σε ελέγξουμε καλύτερα. Την 33. Ψηφίσατε. 30 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. 34. Με γλωσσική διόρθωση, την οποία δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 34 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35, υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Συμβιβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Όχι καταπίπτει 54. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 74. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Σας παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Τροπολογία 76. Σας παρακαλώ να φαίνεστε όταν ψηφίζετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Α, όχι, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει. Πού είμαστε. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τροπολογία 80 έχει αλλάξει μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 80 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Όχι 88, 88, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 92 και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 47 ε, υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Und wir sind wieder in der Zeit. Μάλιστα, προλάβαμε, προλάβαμε. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης, δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να μιλήσετε, έξω από την αίθουσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ, το, 2007 και 2014. Η Μάριαν Χάρκιν είναι η συγγήτρια. Θα συζητήσουμε σήμερα τις τροπολογίες και δίνω αμέσως το λόγο στη Μάριαν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Έχουμε 163 διαχειρίσιμους αριθμούς. Δεν θα ήθελα να διατρέξω τις τροπολογίες μεμονωμένα, γιατί δεν έχουμε χρόνο θα τις ομαδοποιήσω και θα κάνω ορισμένα σχόλια για τις τροπολογίες. Θα ήθελα να πω, μάλλον περισσότερο να ακούσω αυτά που έχουν να πούν οι άλλοι. να μου επεξηγήσουν γιατί τις έχουν ε, υποβάλει. Δηλαδή υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες προτρέχοντας κάπως την ανάγκη αναδιάρθρωσης. Αυτή η συζήτηση έγινε όταν αναθεωρήσαμε το Ταμείο την προηγούμενη φορά. Ε, δηλαδή στο νέο κανονισμό προβλέπεται κάτι τέτοιο, αλλά επειδή ο κανονισμός αφορά τους απολυμένους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε κάπως να προτρέξουμε ως προς την αναδιάρθρωση, κάτι το οποίο είναι θετικό αυτό. Ε, δηλαδή να διαχειριστούμε τις αλλαγές και να προβλέψουμε τις απώλειες και να τις αποτρέψουμε, το Ταμείο Αντιμετώπισης ε, της Παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα ήθελα να πείτε εσείς αν νομίζετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά όσο έχει δεν μπορεί. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η πτυχή του θέματος. Υπήρχαν ορισμένες θετικές τροπολογίες ε, για την αξία των ε, συνεταιρισμών και τον ε, τομέα του εμπορίου γενικότερα. Γιατί το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φύλλο έτσι ώστε η Επιτροπή να μας πει ότι θα γίνουν τόσες απολύσεις, αλλά το Ταμείο Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης μπορεί να το αντιμετωπίσει. Όμως υπήρχε Υπήρχαν ε, τροπολογίες για εμπορικές ως προς εμπορικές συμφωνίες που δεν θα έπρεπε να ενταχθούν εδώ, κατά τη γνώμη μου. Πολύ λεπτομερείς πολλές από αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι το σωστό σημείο για να μιλήσετε υπέρ ή κατά της TTIP και όλων των συμφωνιών που έχουμε με την Αμερική, με τη Ρωσία και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ενταχθούν εδώ, ενώ επιμέρους σημεία μπορούν να ενταχθούν. Αρκετές τροπολογίες υπάρχουν για τη βελτίωση του κανονισμού, ιδιαίτερα για τη διαφάνεια. Θα τις υποστηρίξω. Άλλες ασχολούνται με τις ΜΜΕ και πώς μπορούν να ευεργετηθούν οι εργαζόμενοι δηλαδή στις ΜΜΕ από το Ταμείο Προσαρμογής, ιδιαίτερα στον κοινωνικό διάλογο και την εφαρμογή των μέτρων. Μία από τις τροπολογίες αφορά τις ανασυντάξει νομίζω ότι αφορούν ε, μία τροπολογία του κυρίου Σάντερ να μου επεξηγηθεί όμως σας παρακαλώ. Μιλάμε για μείωση του αριθμού από 500 σε 200. Δεν αντιτίθεμε από πλευράς αρχής, αλλά αυτή η συζήτηση είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι υπάρχει μία εξαίρεση σύμφωνα με την οποία ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ένα 15-16% των ε, αιτήσεων που αφορούν αριθμό πολύ κατώτερο των 500. Αυτό το μέσο ήδη υπάρχει ως προς τον αριθμό των εργαζομένων και λειτουργεί πολύ καλά. Δεν το χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη Άρα η αλλαγή του κανονισμού δεν θα αποτελέσει τη θέμενη αξία. Γνωρίζω από την προηγούμενη φορά ότι θεώρησαν πολλοί ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός, ενώ άλλοι αντιτάχθηκαν στεναρά. Εγώ έχω την άποψη ότι επειδή υπάρχει έτσι και αλλιώς η εξαίρεση από πλευράς κρατών μελών, τότε το θέμα ε, καλύπτεται, γιατί βλέπουμε από τον αριθμό αιτήσεων σε σχέση με τους απολυμμένους, σε σχέση με τις έγκαιρες παρεμβάσεις, τις απολύσεις, τις ε, αντιρρήσεις. Το ίδιο το Ταμείο Προσαρμογής στην ουσία ασχολείται με αυτή την ε, περιστολή και ίσως θα μπορούσατε να υποβάλλετε συγκεκριμένες υποδείξεις για το πώς μπορούμε να καλύψουμε χρόνο. Επίσης υπάρχουν θετικές τροπολογίες για την κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς και σε σχέση με την εξαίρεση, σε σχέση με συγκεκριμένες ανάγκες, ζητώντας και την ε, συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Μιλήσαμε για ένα ποσοστό 32% ως προσετήσεις που γίνονται αποδεκτές και νομίζω ότι θα υπάρξει ευελιξία ανάλογα με τις αιτήσει ως προς τις συγκεκριμένες ανάγκες έτσι ώστε να εμπλακούν οι σωστοί οργανισμοί, οι κατάλληλοι οργανισμοί. Δηλαδή υπάρχει ευελιξία στα κρατημέλη, αλλά και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. Δυστυχώς δύο-τρεις συνάδελφοι ε, ήθελαν να απαλείψουμε την παράγραφο σε σχέση με την ε, εκ νέου απασχόληση. Στα πλαίσια της απασχολησιμότητας όμως, οι πολίτες θεωρούν ότι μπορούν να αναζητήσουν μία εργασία και ιδιαίτερα αν δείτε τις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί πολλοί δεν απασχολήθηκαν καν στο παρελθόν. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ορισμένες τροπολογίες σχετίζονται με το θέμα της τρέχουσας απασχόλησης σε σχέση με την προγενέστρη και αυτό δέχομαι να το συζητήσω. Η οροφή, η δυνάμη του 7β, ε, οδήγησε σε σωρία τροπολογιών θελήσαμε, δώσαμε μεγάλη μάχη για να μειώσουμε την οροφή με σχετική επιτυχία. Και εγώ θα ήθελα να μειώσουμε αυτή την οροφή περαιτέρω, αλλά στις διαβουλεύσεις ως προς την έκθεση αυτή, το μήνυμα που έλαβα στις διαβουλεύσεις ήταν να μην αγγίξουμε αυτή την οροφή γιατί δίνει ευελιξία στους εργαζόμενους. Σήμερα είδαμε ότι στην περίπτωση του Βελγίου γίνεται χρήση ενός 5% για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους ως προς τα επιδόματα κινητικότητας. Δίνει δηλαδή ένα μικρό κίνητρο στους εργαζόμενους και κατά τις διαβουλεύσεις έλαβα και το αντίθετο μήνυμα όπου έγινε λόγος για περιορισμένη χρηματοδότηση του Ταμείου Προσαρμογής. Αυτά ήταν τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αν έχετε ειδικέ τροπολογίες, να μου δώσετε και επεξηγήσεις ε, γιατί τις προωθείτε. Νομίζω όμως ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ε, σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Χάρκιν. Έχουν το λόγο τώρα οι σκιώδεις εισηγητές. Ο Τσάμπα Σόγκορ για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Και εγώ χαίρομαι που είχαμε αρκετές τροπολογίες στην έκθεση. Αυτό καταδεικνύει και πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα λόγω της ε, παγκόσμιας κρίσης ε, που σχετίζεται με τις απολύσεις αλλά και τις διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν στα θέματα αυτά. Κάποιες από τις ε, τροπολογίες είναι θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή, αλλά υπάρχουν και αρκετές τροπολογίες οι οποίες θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της έκθεσης. Κυρίως τροπολογίες που αφορούν που έχει κάνει η ίδια η συγγήτρια για την ε, αξιολόγηση και τη συμμετοχή της τοπικής αγορής εργασίας για να υπάρχει ε, ταχεία επανένταξη απολυμένων εργαζομένων και το να υπάρχει και ε, κατάλληλο ε, ποσοστό ωφέλους, ε, να υπάρχουν προγράμματα στον ε, μεταποιητικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα και την ανάγκη να έχουμε ε, πρόσβαση σε περισσότερους ανέργους και να μπορέσουν να εργαστούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσβλέπω στη συζήτηση με την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για τις συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίτα Ούλφσκοκ για τους σοσιαλδημοκράτες. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν ε, για το έργο της, ε, για την πολύ διεξοδική συνεισφορά της, ε, καθώς επίσης και όλους τους κοιόδης συγητές για τις πάρα πολύ καλές τροπολογίες. Προσβλέπω στη συνεργασία μας και πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει ότι όλοι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ε, το ρόλο του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να υποστηρίξουμε τις βασικές του λειτουργίες ε, και τη μελλοντική του βελτίωση. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει σύμπτωση απόψεων πολλών πολιτικών ομάδων επ' αυτού. Οι τροπολογίες μας από πλευράς σοσιαλδημοκρατών καλύπτουν το θέμα το οποίο αναφέραμε στην αρχική συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή. Είχαμε αναφερθεί ε, στο θέμα των ε, εμπορικών ε, συμφωνιών που πολλές φορές δημιουργούν περιττές καταστάσεις που χρειάζονται υποστήριξη από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να είναι λύση για τις θέσεις εργασίας που χάνονται λόγω κακών εμπορικών συμφωνιών. Δεν αφορά το εμπόριο το θέμα αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργούμε προβλήματα αφενός με το ένα χέρι και από την άλλη να προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα με το άλλο. Καταρχά, το Ταμείο Προσαρμογή στο Παγκοσμιοποίηση έχει περιορισμένα κονδύλια για το ρόλο που έχει να διαδραματίσει, γι' αυτό και κάνουμε έκκληση για περαιτέρω χρηματοδότηση του Ταμείου. Αλλά επίσης ε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιούμε το Ταμείο Προσαρμογής για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Όπως για παράδειγμα ε, περιπτώσεις στις οποίες πλήττεται ένας ολόκληρος τομέας και χρειάζεται μεταρρύθμιση. Πρέπει να υποστηρίξουμε διαρθρωτικές προσαρμογές και όχι ε, κάθε επιχείρηση η οποία αποχωρεί από την Ευρώπη. Και επίση έχουμε υποβάλει και μια τροπολογία για Ευρωπαϊκού κανόνες για την αναδιάρθρωση που να είναι νομική, νομικά δεσμευτική. Ε, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το συμπεριλάβει αυτό επανειλημμένος και θεωρούμε ότι ήγηκε η ώρα να το υλοποιήσουμε. Και πάλι επαναλαμβάνω, το Ταμείο Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση υποτίθεται ότι είναι για κατεπίγουσε περιπτώσει. Δεν είναι ένα ε, ταμείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά για λάθος λόγους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν ε, την ευθύνη των πράξεών τους. Επίσης, ε, θέλουμε να τονίσουμε ότι θέλουμε καλύτερη εποπτεία των συνεπειών ε, των κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογής της παγκοσμιοποίησης ε, μέσω του Eurofonds και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Εάν θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση, πρέπει να χρηματοδοτούνται καταλήλως και εγκαίρως. Σας ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, κυρία Χάρκιν. Και υποστηρίζουμε τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κρασνοδεύσκη για του CCR. Λείπει. Θα ήθελε κάποιο να μιλήσει εκ μέρου του. Όχι. Λιν Μπόιλεν τότε, η επόμενη μιλήτρια για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της στο σχέδιο έκθεσης. Θα αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες που έχουμε υποβάλει ε, οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία εφαρμογής ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ιρλανδία και ε, διαβουλεύσεις με διάφορους ενδιαφερομένους στην Ιρλανδία. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε δει να προκύπτει είναι η έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των προγραμμάτων του Ταμείου Προσαρμογής, το οποίο οδήγησε σε επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ ε, στο Ταμείο και επομένως ε, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι που χρειάζονταν αυτή τη στήριξη δεν την έλαβαν. Για παράδειγμα, η πρόσφατη Lufthansa Technic. Ε, από ό,τι φαίνεται, 1,5 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια του Ταμείου θα επιστραφούν μέχρι το Σεπτέμβριο. Και αυτό το θέμα δεν ήταν δημοσίως γνωστό, ε, ήταν ένα θέμα το οποίο σχετιζόταν με, την, ε, με αίτημα για την ελευθερία στην ε, πληροφόρηση. Επίσης, υπέβαλα κάποιες τροπολογίες που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, φροντίσουν τα κράτη-μέλη να έχουν έναν αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή των προγραμμάτων σε επίπεδο κρατών μελών και αυτοί οι φορείς, αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες ε, ε, δεξιότητες ώστε να διασφαλίσουν ότι θα δαπανώνται στο έπακρο τα κονδύλια τα οποία διατέθονται και θα λογοδοτούν και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη θέλουμε να υπάρχουν εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεωτικά και να περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες για τις εκτιμόμενες δαπάνες και μία επιπλέον αίτηση για έγκριση ώστε να μην υπάρχουν ε, των κονδυλίων. Επίσης, ζητάμε δημοσιοποίηση του περιεχομένου ε, και των συμπερασμάτων της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης και επίσης ε, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη λογοδοσία και πάλι και διαφάνεια. Ε, χαιρόμαστε που παρατείνεται η περίοδος παρέμβασης στα δύο χρόνια και επίση προτείνουμε και μια τροπολογία που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για προγράμματα ε, στα δύο χρόνια από τη στιγμή έγκριση και όχι στα δύο χρόνια από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση. Αυτό προέκυψε από τη διαβούλευση με του ενδιαφερομένου, από την εμπειρία του με την εφαρμογή του Ταμείου. Επίση, εξετάζουμε το θέμα τη ε, κατάρτιση. Το γεγονό ότι πολλά από τα μαθήματα είναι ε, πολυετή προγράμματα, τριετή για παράδειγμα, και μπορεί κάποιο να σταματήσει στα μισά την ε, επιμορφωσή του. Ε, και πρέπει να διασφαλίσουμε, λόγω έλλειψη χρηματοδότηση, πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν την επιμόρφωσή τους και να την ολοκληρώνουν. Ε, κάτι άλλο το οποίο σημειώσαμε ήταν το γεγονός ότι ε, δεν υπήρχε στήριξη από επιλέξιμες επιχειρήσεις και ζητήσαμε ε, ο τομέας του εθελοντισμού και κυρίως μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, να εκπροσωπούνται καταλήλως στο στάδιο του προγραμματισμού γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα αυξήσει την πρόσβαση στις κατάλληλες ανάγκες γιατί θα έχουν εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που χρήζουν ανάγκης και βοήθειας και επομένως ε, θα ε, πηγαίνουμε απευθείας σε αυτούς. Ε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποτανθούν σε οποιοδήποτε οργανισμό ή υπηρεσία θεωρούν ότι χρειάζεται βοήθεια. Επίσης, τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν προβλήματα ε, ως προς την ανεξάρτητη έκθεση της εφαρμογής ε, του προγράμματος μέχρι τώρα και κυρίως ε, επειδή πρέπει να επικεντρωθούν και στο θέμα της ανάγκης συμμετοχής. Πρέπει λοιπόν να δαπανίσουν περαιτέρω κονδύλια για να αποδείξουν ότι όντως υπήρχε συμμετοχή. Είπε κάποια συνάδελφος ότι έχουμε περιορισμένα κονδύλια, επομένως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι γίνεται είναι αποτελεσματικό αποτελεσματικό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεκτείνει την περίοδο στην οποία ε, είναι επιλέξιμη κάποιοι για την στήριξη μέχρι το πλήρη κύκλο των προγραμμάτων ε, ε, του Ταμείου. Αυτά προτείναμε λοιπόν από πλευράς ομάδος και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Στανόκα. Ε, μιλώ εξ ονόντος της κυρίας Μόνικα Βάνα, η οποία ζητά συγγνώμη γιατί έπρεπε να είναι στους συντελνιστές άλλης επιτροπής. Λοιπόν, τα βασικά σημεία της ομάδας μας. Συμφωνούμε με την εισήγηση, με την εισηγήτητρια σε σχέση με τη μείωση του κατοφλίου. Το άρθρο 4 σημείο 2 ε, μιλά για τις ανάγκες ευελιξίας. Το βασικό μας μέλημα, το οποίο αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες, αφορά το γεγονός ότι μερικές χώρες χρησιμοποιούν το Ταμείο Προσαρμογής για τη συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτή τη δυνατότητα. Όταν μιλάμε για επιδόματα, θα πρέπει να μειώσουμε το μερίδιο αυτό σε σχέση και με το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε το Ταμείο Προσαρμογής να προβλέπει μια προστιθέμενη αξία σε οποιοδήποτε κίνηση. Έχουμε υποβάλει 16 τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η, από το EFTD η Λαουρα Τζέα δεν είναι εδώ. Η κυρία Πιτζότα έχει το λόγο. Ο κύριος, με συγχωρείτε. Ε, μάλλον ο αντικαταστάτης λέει «Ζητώ συγγνώμη που η κυρία Μπιτζότο δεν είναι ε, παρούσα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χάρκιν για την εργασία της τα στοιχεία ε, δεν ε, επαρκούν, τα ε, στοιχεία που έχουμε για τους αντικτύπους δεν είναι επαρκή, για αυτό το Ταμείο Προσαρμογής και οι ΜΜΕ δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Τι λέει η κυρία Μπιτζότο, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ τις παρεμβάσεις των συναδέλφων έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία σκιαγράφηση της κατάστασης σε σχέση με τη δράση του Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση του παρελθόντος και τι πρέπει να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Το Ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο, ένα μέσο επίγουσας ανάγκης για να βοηθήσει τους πολίτες όταν χάνουν την εργασία τους μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και της παγκοσμιοποίησης. Ε, ευχαριστώ του συναδέλφους για τις ανάγκες ε, του Ταμείου, όπως τις όρισαν, μέσα στα πλαίσια της λιτότητας που όρισε η Τρόικα, κάτι το οποίο οδήγησε σε μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και εξωτερήκευση ή εξωτερική ανάθεση έργων. Συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι η οικονομική κρίση έχει μεγαλύτερη επίπτωση στις ΜΜΕ με λιγότερο από 500 εργαζόμενους, γι' αυτό θα πρέπει να μειώσουμε το κατόφλι απολύσεων για να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση. Το Ταμείο δεν επιλύει το θέμα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε το Ταμείο Προσαρμογής να μην αποτελέσει πανάκια για την σύσταση και ε, ε, έγκριση συμφωνιών όπως το TIP, όπου ε, και σύμφωνα με το οποίο χάνονται τουλάχιστον 600.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε ότι το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα κείμενα σε σχέση με τις επισκέψεις επιθεώρησης. Σας ευχαριστώ που την ακούσατε μέσω εμού. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε τώρα ο γύρος των σχεδόν εισηγητών. Τώρα θα θέσω το λόγο στην κυρία Άγνες Ιονκέριους. Ναι, και είπα και εγώ να πάρω την ευκαιρία να παρευρεθώ και στη συνεδρίαση της ε, ΙΝΤΑ και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στην έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, διότι και εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις και νομίζω πως θα μπορούσαν αυτές οι λύσεις να βοηθήσουν και τη Μάριαν Χάρκινγκ σε αυτό που ε, προσπαθεί να κάνει τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη δουλειά σας, αλλά αφήστε με να πω το εξής να σας εκθέσω την άποψη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ για την παγκοσμιοποίηση. Όπως είπε ήδη η κυρία Ουλσκοκ, δεν είναι αυτή η ευκαιρία για να τοποθετηθούμε κατά των εμπορικών συμφωνιών. Ούτε είναι και ο τρόπος να διορθώσουμε μια κακή συμφωνία. Στην Επιτροπή Ίντα ζητούμε ε, σωστές εμπορικές συμφωνίες. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και μια πάρα πολύ καλή εμπορική συμφωνία θα έχει νικητές και χαμένους. Και φυσικά όταν δουλέψει κανείς ε, καλά, οι νικητές θα είναι περισσότεροι από τους ιτημένους. αλλά και οι πολίτες που εργάζονται σε τομείς που θεωρούνται παραδοσιακά χαμένοι και αυτοί θα μπορούν να βρουν βοήθεια για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Και πολύ συχνά μάλιστα, αντί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από την πλευρά των τομέων που πάσχουν ή των περιοχών που πάσχουν, που υστερούν, πολλές φορές ε, εστιάζουμε στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν γίνεται δηλαδή μία ε, συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα βοηθήσουμε εκείνους τους εργαζόμενους, εκείνες τις εταιρείες, τις περιφερειές που έχουν ανάγκη. Και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ προσπαθήσαμε να ζητήσουμε ε, εκτός, ε, εκτιμήσεις αντικτύπου προτού γίνουν προτάσεις και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την δημόσια διαβούλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ ζητάμε κάποιο εθνικό κοινωνικό σχέδιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου εργαζόμενοι και εργοδότες θα ε, συζητούν μαζί και θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα εγκαίρως παρά ε, όταν η ανεργία θα έχει ήδη φτάσει υψηλά ποσοστά. Και επίσης ζητούμε να χαμηλώσει το κατόφλι για την επιλεξιμότητα στο Ταμείο. Αν θέλουμε πραγματικά να στείλουμε ένα μήνυμα, πρέπει να είμαστε στο πλευρό και των χαμένων από αυτή την ε, μεγάλη μάχη που έχει προκαλέσει η παγκοσμιοποίηση. Και είναι σημαντικό πιστεύω να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Γνωρίζω για τη δυνατότητα παρεκκλήσεων που υπάρχει, όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία δήλωση, να τοποθετηθούμε εδώ. Επίσης, είπαμε και για τα TDI στα εμπορικά μέσα άμυνας. Μιλάμε επίσης και για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας, για τον κοινωνικό διάλογο, εκτιμήσεις αντικτύπου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτά λοιπόν αναφέρουμε στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, αυτά ζητάμε και ελπίζω και εσείς να τα συμπεριλάβετε στην εκθεσή σας. Επίσης να σας πω ότι αν μπορώ να βοηθήσω με διευκρινήσεις ή οτιδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Ρένα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Μαριάν Χάρκιν για τα όσα κάνει ήδη σε επίπεδο Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και για την έκθεση και την ε, Μαρίτα για τα όσα έχει κάνει και αυτή. Ε, νομίζω ότι βρίσκομαι στην ίδια θέση με τη συνάδελφο που μόλις μίλησε. Και εγώ είμαι μέλος και της ΣΥΝΤΑ και της Επιτροπής Απασχόλησης. Επομένως πρέπει ε, να δούμε και τι γίνεται με τη χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογής στην κατά ε, παγκοσμιοποίηση και των εμπορικών συμφωνιών που προσπαθεί να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν ε, εις βάθος μελέτες επιπτώσεων και σε περιφερειακά και σε τομεακά ζητήματα για τις διάφορες αλλαγές, διότι όπως είπε και η συνάδελφος, ακόμα και στις καλύτερες εμπορικές συμφωνίες, πάντα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι οι σε κάποιους τομείς και σε κάποιες περιοχές, επομένως πρέπει αυτές οι συμφωνίες να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα στοιχεία. Ε, πρέπει να προσέξουμε όμως κάτι κυρίως όσον αφορά τα ταμεία και τις ε, περιοχές ε, που πλήττονται. Όταν υπάρχει μια διαδοχή τομεακής αναδιάρθρωσης που επικεντρώνεται σε μια περιοχή, βλέπουμε ορισμένες φορές και απερίμωση αυτών των περιοχών, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακατευθύνουμε αυτούς τους εργαζομένους, γιατί δεν υπάρχει ένας κλάδος πια, έχει καταστραφεί. Επομένως, οι δυνατότητες δημιουργίας αυτοαπασχόλησης για να παραμείνουμε σε, στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια περιοχή, μου φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το υποστηρίξουμε και μάλιστα περισσότερο από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Διότι πρέπει να φροντίσουμε οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να μην χάσουν τις δραστηριότητές τους και τον πληθυσμό τους. Επομένως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο το σημείο αυτό. Κάτι ακόμα ως προς το Ταμείο, το οποίο σχεδίζεται πάντα με το θέμα της επανένταξης. Είπαμε ότι Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και των διαφόρων κλάδων, αλλά ε, και πάλι σε κάποιες ε, ε, περιοχές που είναι περιοχές υψηλού ποσοστού ανεργίας δεν δίνεται απόλυτα η δυνατότητα αυτών των ε, ε, ανθρώπων που έχουν και χαμηλά προσόντα να αλλάξουν κλάδο. Πρέπει να τις προσέξουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα για να καλύψουν αυτές τους μακροχρόνια ανέργους και επίσης να δούμε και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν και τόσο πολλά προσόντα. Υπάρχουν και άλλα ταμεία βέβαια που ρυθμίζουν κάποια προβλήματα, για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τους στόχους του κάθε ταμείου. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση, που έχει συγκεκριμένα ε, κονδύλια, να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να υπάρχει ένταξη στην αγορά εργασία. Υπάρχουν και άλλα ταμεία, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΦΕΝΤΕΡ, το Γεωργικό Ταμείο, που μπορούν να βοηθήσουν αυτού του ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση, αφού έλαβαν το λόγο όλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Τζίλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το λόγο και αφήστε με να αρχίσω αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής για την δουλειά που έχετε κάνει και την προσοχή που έχετε δώσει στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Από πλευράς Επιτροπής θα ήθελα να κάνω κάποια γενικότερα σχόλια ως αντίδραση αυτό, σε αυτά που άκουσα, ε, όχι σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά γενικά. Όπως και η κυρία Χάρκιν, θα αρχίσω και εγώ από το ίδιο, η αναμονή για την αναρδιάρθρωση δεν είναι ε, βασικό στοιχείο, δεν είναι ο ρόλος του Ταμείου. Η, προσ... η πρόβλεψη μάλλον, με συγχωρείτε. Το Ταμείο δεν είναι σε θέση να προβλέπει ούτε σε αυτή τη μορφή που έχει τώρα, ούτε στο μέλλον της επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών. Στη μορφή που έχει τώρα, το Ταμείο δεν έχει προσανατολισμό σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, τι μπορεί να κάνει ήδη από τώρα η Επιτροπή. Πιστεύω πως μπορούμε να επωφεληθούμε αμοιβαία, να δούμε δηλαδή ε, τα στοιχεία από τις εθνικές ε, αρχές μια φορά το χρόνο και να διευκολύνουμε μια αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για όλους τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από τα διάφορα κράτη-μέλη και να ανταλλάξουμε εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες ε, με τα μέλη τα οποία δεν είχαν δείξει τόσο μεγάλη επιτυχία. Και εδώ πιστεύω πως η καλύτερη εφαρμογή είναι βασική λέξη. Η εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επίσης ε, η κερία σημασίας. Πρέπει να ε, εστιάσουμε εκεί έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Να μην ξεχάσω επίσης να αναφέρω ότι μία από τις συστάσεις που αφορούν το θέμα αυτό είναι ε, η έκκληση για, καλύτερη, για καλύτερο έλεγχο. Περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ε, φορείς, περισσότερες εθνικές αρχές θα πληροφορηθούν, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το Ταμείο και για τη χρήση του. Και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά και την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές για τα σχόλια και τις προτάσεις τους και σίγουρα θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όσα είπατε και θα λάβετε ένα συμφαστικό κείμενο από εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Μαριαν Χάρκινγκ για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ όλους που λάβατε το λόγο, τους Σκιώδης και άλλους ομιλητές. Ε, δέχομαι τη δική σας θεώρηση των πραγμάτων, την εκτιμώ. Συμφωνώ σε σχέση με τον ε, συγκεντρωτισμό που υπάρχει σε ορισμένους τομείς, όπως είπε ο κύριος Σόγκαρ, και υπάρχουν και πολύ καλές τροπολογίες σε σχέση με την προστασία του πλαισίου. Ως προς τις ε, εμπορικές συμφωνίες, συμφωνώ με την κυρία Ολσκοκ ότι δεν θα, πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα προσπαθώντας να λύσουμε εν μέρη, να επιλύσουμε εν μέρη την κατάσταση. Καθίσταται σαφές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν ότι το Ταμείο χρησιμοποιείται ως φίλος οικής, έτσι ώστε ο Επίτροπος Εμπορίου να πει ότι ναι, υπάρχουν απολύσεις, αλλά έχουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σαν να πρόκειται για ε, πανάκια. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια ετησίως απώλειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα, δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί το Ταμείο αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε λανθασμένες πολιτικές δηλώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει με μια εμπορική συμφωνία, θα υπάρξουν απώλειες, αλλά έχουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι μια λανθασμένη πολιτική δήλωση. Συμφωνώ με την κυρία Ολσκοκ σε σχέση με τις διαρθρωτικές προσαρμογές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει λεπτομεριακή συζήτηση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες προτάσεις να υποβάλουμε. Και φυσικά αυτή η έκθεση οδηγεί και σε πολιτικές δηλώσεις. Πρόκειται για ένα ταμείο Τεπίγουσας ανάγκης. Η Λιν μίλησε για ανεπαρκή δαπάνη, αλλά πολλές φορές έχουμε υπολοιματικά ε, ποσά, γιατί γίνεται επαναπρόσληψη, δηλαδή ε, μπορεί να υπάρχει και επαναπρόσληψη και κατάρτιση, γι' αυτό υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. θα πρέπει να υπάρξει μία ενδιάμεση, ενδιάμεση αποτίμηση λειτουργίας του Ταμείου Προσαρμογής. Να δούμε δηλαδή τι πρόοδος έχει επιτελεστεί και κατά πόσο μπορούν να δαπανηθούν τα χρήματα που ζήτησαν για αυτούς που έχουν πρόσβαση. Δεν πρέπει να αποστέλλονται πίσω τα χρήματα, διότι ε, δυστυχώς η ελληματική δαπάνη ανέρχεται σε 50% για θετικούς ή αρνητικούς λόγους. Θα πρέπει να διακρίνουμε τους μεν από τους δε. Πιστεύω σε σχέση ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο οργανισμός αναπροσαρμογής για τα τρία χρόνια έδωσα και εγώ μια μεγάλη μάχη στη τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου. Δεν με υποστήριξαν οι συνάδελφοι γιατί είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν να προβάλλουν μια κατάρτιση τουλάχιστον ε, τριετή. Μιλήσαμε όμως ε, για ένα ταμείο επίγουσας ανάγκης και ίσως αυτό το θέμα θα πρέπει να το δει το ΕΚΤΑ δέχομαι την εξαίρεση για τις ε, ανάγκες που θα ανακύψουν πέρα από το 2017. Η κυρία Βάνα μίλησε για το 7β, το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να μας απασχολήσει και ελπίζω να επέλθει συμφωνία. Η κυρία Μπιτζότο μίλησε για τις ΜΜΕ, αυτό είναι πολύ σημαντικό και η μείωση του κατοφλίου είναι σημαντική. Εγώ δεν αντιτίθεμαι, αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο θα βελτιώσει τον κανονισμό. Δέχομαι τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Το συζήτησα με την Κομισιόν, αλλά εάν δεν δημοσιοποιούν τα κράτη-μέλη τα έγγραφα, τότε δεν μπορεί να επιληθεί τίποτα. Σας ευχαριστώ ε, για τη συνεισφορά σας από την ίντα. Δύο σημαντικά ζητήματα ετέθησαν. Το ένα αφορά το γεγονός ότι σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Θα πρέπει να ε, κάνουμε μια αποτίμηση γιατί μιλάμε για τομείς, για περιφέρειες και οι περιφέρειες ε, έχουν εξαλειφθεί από τον χάρτη. Μιλάμε για 600.000 απώλειες και μπορεί κανείς να μετακινηθεί από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Δεν σημαίνει ότι θα βρει νέα εργασία. Υπάρχουν επιπτώσεις σε τομείς και περιφέρειες. Χρειάζεται μια καλύτερη αξιολόγηση. Εάν υπάρχει κοινωνικός διάλογος, ε, τότε μπορεί κανείς να διαχειριστεί το εμπόριο. Μερικοί δεν το θέλουν καν, ας το πούν ανοιχτά. Εάν το υποστηρίζετε όμως, θα πρέπει να προωθήσετε προτάσεις που εξασφαλίζουν ε, την καλύτερη έκβαση η σωστή αξιολόγηση μαζί με τον κοινωνικό διάλογο μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Ρένα μίλησε για περιφέρειες και μπορούμε να προσθέσουμε κάτι και σε αυτό. Το Ταμείο δεν είναι πανάκια. Άκουσα τι είπε η Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με την αναδιάρθρωση το Ταμείο αλλά πρέπει να κάνουμε μία πολιτική δήλωση ως προς τη σημασία αυτού. Υποστηρίζω το έργο της Κομισιόν να υπάρξει μία αμοιβαία κατάρτιση, τα κράτη-μέλη να μάθουν τα μεν από τα δε. Αυτή είναι μια γενική αποτίμηση αυτών που άκουσα. Χαίρομαι διότι η ευρεία πλειοψηφία προβάλλει θετικά σημεία να βελτιώσουμε δηλαδή τον κανονισμό και να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα διεξαχθεί στις 15 ή 16 Ιουνίου. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και εύχομαι σε όλους τους σκιώδες συζητητές και όλους τους καλή δουλειά και καλά αποτελέσματα. Εμείς θα τα πούμε στις 30 Μαΐου στις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Όχι 3 με 6.30 αλλά 3,5 με 7. Σας εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ και καλή συνέχεια.